Okay, we should start. Αρχίζουμε παρακαλώ. Σας καλωσορίζω με μία μικρή καθυστέρηση στη συνεδρίασή μας. περιμέναμε να έρθουν περισσότεροι. Ξεκινάμε. Όπως ξέρετε, χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια ακρόαση. Από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και για πρώτη φορά εφαρμόσαμε αυτή, αυτή, αυτό το νέο σύστημα. Δηλαδή, δύο επιτροπές συναρμόδιες σε ίδιο επίπεδο για το ίδιο θέμα. Πήγε πολύ καλά. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω, οπότε την εγκρίνουμε. Έγκριση των πρακτικών τώρα. Από τα πρακτικά της 21ης-22ης Ιανουαρίου και 27ης Ιανουαρίου 2015. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4. Ανακοινώσει του Προέδρου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των συντονιστών της 21ης Ιανουαρίου του 2015 με συμφωνία των μελών της Επιτροπής αναθέσαμε στον κύριο Δεκάστρο να εκπονήσει για την Επιτροπή μας ένα σχέδιο ψηφίσματος με θέμα την ε, Διεθνή Έκθεση, την ΕΞΠΟ του Μιλάνου για το 2015. Αυτό το ψήφισμα θα συνοδεύσει την προφορική ερώτηση που έχει ήδη κατατεθεί για την Expo του Μιλάνου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τεκάστρο για να μας εξηγήσει το θέμα και να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Έχετε το λόγο κύριε Δεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ψήφισμα ήδη ετοιμάστηκε και είναι διαθέσιμο στα αγγλικά. Πρόκειται για ένα ψήφισμα που προσπάθησε να ε, συμπεριλάβει τις συζητήσεις που είχαμε στη σειρά των ακροάσεων που κάναμε για το θέμα του Feeding the Planet Energy for Life, που είναι το θέμα τη παγκόσμια έκθεση του 2015. Το ψήφισμα προφανώ θα είναι ένα ψήφισμα της δικής μας Επιτροπής, επιτροπή Γεωργίας, που και ευχόμαστε πέραν των δικών μα εργασιών να μπορέσουν ε, να συμπεριληφθούν και οι θέσει και γνωμοδοτήσει άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται για, για την πολύ σημαντική αυτή παγκόσμια εκδήλωση που θα γίνει από την 1η Μαΐου του 2015. Το ψήφισμα θα μεταφραστεί και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες μεθαύριο, πριν τις 25. Επαναλαμβάνω ότι είναι διαθέσιμο ότι είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και μεθαύριο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Λόγω προβλημάτων χρόνου τώρα και μελετήσαμε όλε τι δυνατότητε, αλλά μπορέσουμε να εγκρίνουμε το ψήφισμα στην Ολομέλεια πριν τα εγγένεια της ΕΞΠΟ έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να υποβάλουμε τροπολογίε. Θα ζητούσε λοιπόν από του συναδέλφου να δουν το ψήφισμα γρήγορα ότι θα υπάρξει πολύ δημόσιο ενδιαφέρον όταν στο Στρασβούργο, ακριβώς λίγες μέρες πριν τα γένεια της έκθεσης, υποβληθεί το ψήφισμα. Η προθεσμία λοιπόν είναι δυστυχώς με Παρασκευή 27 του μηνός. Δύο-τρεις μέρες δηλαδή. Αυτή την Παρασκευή τώρα. Σε τρεις μέρες, τέσσερις. Αν μπορείτε να δουλέψετε αγγλικά υπάρχει το κείμενο όπως σας είπα. Αν χρειάζεστε τη μετάφραση σε δική σας γλώσσα μέχρι τις 25 θα έχετε όλες τις μεταφράσεις. Θα έχετε λοιπόν δύο μέρες μόνο για να μπορέσετε να δείτε το κείμενο. Πάντως ε, συζητήσαμε πολλές φορές το θέμα της παγκόσμιας έκθεσης μεταξύ μας. Θα ευχόμουν να είναι σημαντικό πολιτική συζήτηση, εμείς καθοδηγήσαμε σαν επιτροπή τη συζήτηση, το θέμα της ψητιστικής ασφάλειας, ε, το θέμα της ε, έκθεσης είναι μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εδώ περιλαμβάνονται και άλλες παράμετροι. Έρευνα, σπατάλη, βιώσιμη διαχείριση των ε, φυσικών πόρων είναι θέματα της Επιτροπής μας. Είναι σκόπιμο λοιπόν να μπορέσουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό και η Επιτροπή μας να είναι η ηγέτης Επιτροπή που θα υποβάλει στην Ολομέλεια στο το ψήφισμα. Αυτά. Δεν γίνεται ούτε συζήτηση ούτε παρουσίαση. Μία θερμή πρόσκληση που απευθύνω σε όλους σας, ούτως ώστε να δείτε όλοι το ψήφισμα. Είναι ένα ψήφισμα που εμπλέκει όλες τις πολιτικές ομάδες και την Επιτροπή μας συνολικά. Νομίζω ότι τα είπα όλα τροπολογίες προθεσμία 27 Δευτέρου. Το κείμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες στι 25, ενώ ήδη είναι διαθέσιμο στα αγγλικά σήμερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Όντως το θέμα αυτό το εξετάσαμε πολλές φορές ε, στην Επιτροπή μας και δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχο. και πιστεύω ότι θα διεκπαιρεώσουμε τη διαδικασία αυτή χωρίς πρόβλημα. Θα συνεχίσει ο κύριος Ντεκάστρο να είναι ο αρμόδιος και θα χειριστεί τη συζήτηση και την διαμόρφωση, την οριστική του ψηφίσματος. Ενημερωθήκαμε και για τις προθεσμίες κατάθεσης των τροπολογιών, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε εγκαίρως το ψήφισμα στην Ολομέλεια. Όπως είπε και ο κύριος Δεκάστρο, εμείς είμαστε η καθήλια αρμόδια επιτροπή γι' αυτό. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει διερμηνία σε 20 γλώσσες με εξαίρεση εστονικά, μαλτέζικα και σλοβακικά. Έχει έρθει στο μεταξύ και ο επόμενος μας εισηγητής, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ο τομέας των απορροκυπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Θα εξετάσουμε λοιπόν ε, την έκθεση του κυρίου Μέλο που πραγματεύεται την κατάσταση στην αγορά προκυπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις, οργανώσει οργανώσεις παραγωγών και τα επιχειρησιακά προγράμματα που διαχειρίζονται. Ε, ξέρετε, το θέμα, δεν υπάρχει αρκετή οργάνωση, ιδιαίτερα στις νέες χώρες. Είναι σημαντική η οργάνωση σε ενώσεις, οργανώσεις παραγωγών για τη διαχείριση του τομέα και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται και κάποιες παρεμβάσεις. Στις 22 Ιανουαρίου, θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε διοργανώσει και ένα σεμινάριο, ένα εργαστήριο με θέμα τον τομέα των απορκυπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Λάβαμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες και είμαστε πια έτοιμοι για πιο ευρυθή συζήτηση θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Νούνο Μέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να σας πω ότι το σχέδιο ψηφίσμα, το σχέδιο έκθεσης ε, εμπλουτίστηκε με τις ε, παρατηρήσεις πολλών ενδιαφερομένων ε, και οργανώσεων αλλά και ευρωβουλευτών και περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες πτυχές του θέματος. Θα σταθώ σε μερικές από τις πτυχές αυτές. Για παράδειγμα, την ανάγκη να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες οργανώσεις παραγωγών ε, και να στηρίξουμε είτε τη δημιουργία νέων είτε τη συγχώνευση κάποιων οργανώσεων παραγωγών στο μέλλον Επίσης να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των χωρών και την ανάπτυξη των οργανώσεων παραγωγών σε αυτές. Είχαμε μια πολύ καλή έκθεση στην Επίτροπή μας και πολύ καλό σεμινάριο με παρουσίαση των διαφορών ε, των οργανώσεων παραγωγών μεταξύ χωρών του Βορρά και του Νότου. Μερικές φορές δυστυχώς η παραγωγή είναι εχμάλωτη των ε, μεγάλων αλυσίδων διανομής και έχουν ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύ, γι' αυτό και έχει νόημα η οργάνωσή τους σε οργανώσεις. Επίσης, ε, δεν πιστεύουμε στον καπιταλισμό της αγοράς. Δεν ε, θα πρέπει να ισχύει και εδώ η αρχή του ο αυτός ο Πρέπει να βοηθήσουμε του παραγωγού να οργανωθούν για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του ε, δύναμη. Επίση, η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή στι εισαγωγέ, ενώ ορθώνει εμπόδια στι εξαγωγέ. Χρειαζόμαστε και πολιτικέ διαπαιδαγώγηση για την ενίσχυση τη κατανάλωση απορροκυπευτικών. Αναφέρεται το γεγονό ότι πρόκειται για ευαλείωτα αναλώσιμα αγαθά που είναι ευπαθή και που πολλές φορές ε, πλήττονται από κρίσεις όπως ε, ισχύει με το ρωσικό εμπάργο την κρίση στην Ουκρανία. Ε, θα πρέπει να μπορούν οι οργανώσεις ε, παραγωγών να προσλαμβάνουν ικανούς μάνατζερ, διαχειριστές. Γιατί μερικές φορές μπορεί τα μέλη των οργανώσεων παραγωγών να είναι καλοί και άξιοι γεωργοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και επαρκής μάνατζερ για τη διαχείριση προγραμμάτων. Αυτά λοιπόν ε, σε, ήταν εν ολίγης τα σημεία της έκθεσής μου και να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι είμαι ανοιχτός και διαλλακτικός. Περιμένω τις προτάσεις σας και σε συνεργασία και με τους κοιόδης ηγητές των κομμάτων πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε έγγραφο που θα απηχεί τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη συζήτηση. Ζήτησε πρώτα το λόγο η κυρία Γιλέρα. Παρακαλώ κυρία Γιλέρα, έχετε το λόγο. Muchas Eh, Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Πολύ σημαντική έκθεση κύριε Μέλο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ιδιαίτερος για χώρες όπως η Ισπανία και όπως η περιοχή μου, η Ανδαλουσία όπου τα προκυπευτικά παίζουν μεγάλο ρόλο, έχουν μεγάλο βάρος στην γεωργία της περιοχής. Γενικά συμφωνώ με την έκθεσή σας, αλλά να κάνω μερικές ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κατά τη γνώμη μου, η κοινή οργάνωση αγοράς για τα οποροκυπευτικά λειτουργεί καλά σε γενικές γραμμές, αλλά βέβαια χρειάζονται κάποιες ε, βελτιώσεις στο σύστημα που θα βοηθήσουν θα ενισχύσουν τους παραγωγούς, όπως είπατε, γιατί υπάρχει ανισορροπία στην διατροφική αλυσίδα, όχι μόνο για τα οποροκυπευτικά, σε όλους τους τομείς που είναι σε βάρος των παραγωγών. Οπότε χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, κάποια ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών για να μειωθεί αυτή η ανισορροπία στη διατροφική αλυσίδα. Διότι κατά τη γνώμη κάτι δεν λειτουργεί καλά όπως είδαμε, είναι οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων. Όταν πρέπει να παρέμβουμε, διαπιστώνουμε ότι όταν έχουμε σοβαρές κρίσεις όπως η E. και το εμπάργο ε, της Ρωσίας, τότε βλέπουμε ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης ε, κρίσεων δεν λειτουργούν γιατί δεν κάνουμε αποσύρσεις, γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα. Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα κυριότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε και μέσω αυτής της ε, έκθεσης. Να βελτιώσουμε αυτούς τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσης διότι δεν λειτουργούν. Επίσης, είναι αναγκαίο να δώσουμε περισσότερα κίνητρα. Είπατε, για τη δημιουργία αλλά και για τη συγχώνευση και στις ε, ε, βέλτιστες διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι οργανώσεις παραγωγών όπορο-κυπευτικών, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερο βάρος στη διατροφική αλυσίδα. Βεβαίως, να δημιουργούνται, γιατί είναι πολύ άνηση η κατάσταση από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο και υφίστανται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να τις βοηθάμε να δημιουργούνται και να έχουν και μεγαλύτερες διαστάσεις αυτές οι οργανώσεις. Επίσης, να σας πω ότι ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο να δούμε ακριβώς και τις ρυθμιστικές διατάξεις Να υπάρχουν δηλαδή εθνικές ρυθμίσεις, αλλά να υπάρχει και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο μία διεπαγγελματική οργάνωση για να βελτιωθεί η κατάσταση γενικά σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας. Κάτι άλλο, θα υποβάλω μία τροπολογία για να προωθήσω όλα αυτά που είπα, αλλά θέλω να σας συγχαρώ, είναι πολύ καλή έκθεση το αρχικό κείμενο και σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, στο μεταξύ έγινε ιδιαίτερα μακροσκελής ο κατάλογος των ομιλητών, γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε στο 1,5 λεπτό ο καθένας. Γιατί επιμικήθηκε πολύ ο κατάλογος. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους ε, σκιώδεις ηγητές, ο κύριος Χαϊτέμα. Παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. also thank you. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής ε, αποτυπώνει καλά την κατάσταση στον τομέα αυτό. Βλέπετε ότι έχει αυξηθεί το πίπεδο οργάνωση των παραγωγών, αλλά υπάρχουν πολλές και μεγάλες ανισότητες μεταξύ χωρών. Αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας. Αλλά σε κάποιες ε, χώρες μέλη. Είναι πολύ μικρή η παραγωγή και είναι δύσκολο να υπάρξουν οργανώσει. Καλό είναι να το ξέρουμε αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικέ οι οργανώσει παραγωγών, ιδίω σε περίοδου κρίση, όπω είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, για να μπορούν να έχουν ισχυρή θέση στην αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κανόνε ανταγωνισμού πρέπει να είναι σαφέστεροι για του οργανώσει παραγωγών. Και κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελα να σχολιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η νομική ασφάλεια. Για να έχουν τη δυνατότητα να δράσουν, να προσαρμοστούν και να διορθώσουν τα λειτουργικά τους προγράμματα οργανώσεις παραγωγών, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να είναι σαφέστεροι και επίσης να υποβάλλονται ταχύτερα. Ορισμένες φορές θέλει δύο χρόνια η Κομισιόν για να κάνει κάποιους ελέγχους. Επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι, ενώ οι... σύνδεσμοι οι... οργανώσεων παραγωγών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι κανόνες λοιπόν για αυτές τις οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι σαφέστεροι για τους, για τις, για τους συνδέσμους οργανώσεων παραγωγών. Επίσης θα ήθελα να μειωθεί η γραφειοκρατία γιατί πολλές φορές ε, δεν ευνοεί, την, αντίθετα παρεμποδίζει την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να συγχαρώ και εγώ τον ε, εισηγητή κύριο Μέλο για τη δουλειά που έχει κάνει. Η έκθεσή του καλύπτει πολλά θέματα, την οργάνωση του κλάδου, των οπορικευτικών που παραμένει ακόμα προβληματική, υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό σε κάποια κομμάτια τη αλυσίδια τροφή. το πρόβλημα των εργαλείων διαχείριση και πρόληψη των κρίσεων πέραν άλλων ε, ζητημάτων κομβικού χαρακτήρα όπως οι οργανώσεις παραγωγών. Το υφιστάμενο σύστημα προστασίας των απογευτικών που έχουν προτείνει συμβάλλει αλλά δεν επαρκεί για την ορθή λειτουργία του συστήματος όπως προτείνει η εμπειρία. Για παράδειγμα, θα ήταν αναγκαία να υπάρχει μεγαλύτερη απλοποίηση και να υπάρχουν προσαρμογές σε μια σειρά εργαλείων όπως που προβλέπονται για τη διαχείριση των κινδύνων και τελειοποίηση των κινήτων προς τους ε, οργανώσεις, παραγωγών. Είναι γνωστό σε όλου ότι ο βαθμό οργάνωση του κλάδου των οπωροκευτικών είναι χαμηλό σε πολλά κρατημέλη και σε πολλέ περιφέρειε τη Ένωση. Πολλοί παράγοντε ε, περιορίζουν ε, την ομαδοποίηση των οργανώσεων παραγωγών, ιδίω οι σύνθετε διαδικασίε για την αναγνώρισή του από τα κράτη. Ένα δεύτερο σημείο που θα έπρεπε να προβληθεί είναι τα εργαλεία διαχείρισης και πρόληψης των κρίσεων που είναι στη διάθεση των οργανώσεων παραγωγών αυτή τη στιγμή όπως η χρήση πόρων ε, αμοιβαίων κεφαλαίων για την προστασία των παραγωγών που ανακύπτουν, που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των, της τελευταίας κρίσης με το ρωσικό εμπάργο. Εγώ πάω πιο γρήγορα, αλλά πραγματικά, Πρόεδρε, ο χρόνος που μα δίνεται δεν είναι αρκετός. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια δυνατότητα να ε, αναδεικνύουμε τη δουλειά που έχει γίνει. Εγώ βρίσκομαι στη μέση της παρέμβασής μου μόνο, που είναι καρπός μιας δουλειά που έχουμε κάνει πολύ μαζί. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να μα δώσετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τι θέσει μα. Πάω, γρήγορα. Τρίτο, σε κάποια κράτη-μέλη τα επιχειρησιακά προγράμματα συμβάλλουν με σπάνιο ή καθόλου τρόπο στην αύξηση της εμπορικής αξίας των ε, προϊόντων που έχουν προωθηθεί στην αγορά, ε, ενώ συγκεντρώνουν την προσφορά. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε κατά συνέπεια να υποστηρίξουν οργανώσει παραγωγών και να ενισχύσουν τη συμβατική ικανότητά τους, λαμβάνοντα υπόψη την καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς. Εν τέλει θα ήθελα να σταθώ σε κάποιε διαστάσει που μπορούσαν να βελτιώσουν κατά άποψή μου την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο καταρχήν να αναφέρουμε σαφώς ε, τους ε, στόχους κατά προτεραιότητα με ρητή και ποσοτική τοποθέτηση για να μπορέσουμε να δώσουμε με αντικειμενικό τρόπο τα επιτευθέντα αποτελέσματα και σε σχέση με, τους, ε, με τις στρατηγικές και τους στόχους που είχαν τεθεί για να βελτιώσουμε την τη συνολική ανταγωνιστικότητα. Δεύτερο θέμα, να προβλέψουμε καλύτερη ενημέρωση. Αυτό υπογραμμίστηκε και από τον εισηγητή τον ίδιο. Πολύ συχνά το management δεν έχει σωστή κατάρτιση. Και τέλος να προωθήσουμε μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων στόχων. Ευχαριστώ. Σα άφησα λίγο χρόνο παραπάνω γιατί είστε σκιώδης ηγητή. Η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον κύριο Μέλου για την έκθεσή του αντιμετωπίζει τα δύο βασικά θέματα ανησυχίας. Ορισμένες αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές στη διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό έχω εργαστεί και εγώ και θα συνεργαστώ μαζί σας. Το δεύτερο, πόσο περίπλοκη και γραφειοκρατική είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουν οι οργανώσεις παραγωγών. Το 2013 για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια και ορισμένα άλλα μέσα διαχείρισης ε, κρίσεων θα πρέπει να το συζητήσουμε και αύριο όταν θα συζητήσουμε για τις διαφορές μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε ε, για το πώς λειτουργεί το δικό του σύστημα και πώς μπορεί αυτό να μας βοηθήσει. Ε, θα έχω κάποιες τροπολογίες, αλλά θεωρώ ότι είναι θαυμάσια εκθεσή σα και θα μας βοηθήσει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτού του τομέα. Ευχαριστώ κύριε Σεμπάστια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μέλο. Καλή έκθεσή σας και συγχαρητήρια. Μίλησα με συνδικάτα, γεωργικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγών και πολλοί ε, με πένεσαν ε, και μου είπαν να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας. Ενισχύω και τις ε, επικρίσεις που κάνατε και τα σημαντικά προβλήματα που επισημάνατε. Έχουμε εγκατάλειψη γεών, δυστυχώς έχουμε γύρανση των γεωργών. Επισημάνατε όλα αυτά τα προβλήματα, καθώς και τα προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα, με τις εισαγωγέ από τρίτες χώρες και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι από τη Βαλένσια, όπως και οι συνάδελφος από την Ισπανία, και μάλιστα ε, έχουμε μεγάλη παραγωγή φρούτων που κατά παράδοση δρομολογούσαμε προς τη Ρωσία. Μας έπληξε λοιπόν το ρωσικό εμπάργο. Και οι οργανώσεις παραγωγών δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μέσο για τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε αυτές τις ε, ενώσεις αλλά κυρίως για να βοηθήσουν τους γεωργούς. Ενώ οι πωλήσει δεν έχουν βελτιωθεί δυστυχώς. Άρα δεν, ε, δεν επιτυχάνεται ο στόχος μας που ήταν η ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε το μέλλον της γεωργίας. Οπότε αυτό το σύστημα της οργάνωσης παραγωγών δεν ελέγχθηκε σωστά και γι' αυτό δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Μέλλο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Χαίρο που έθεσε τη έμφαση σε κάποιες βασικές αρχές. Για παράδειγμα, η μείωση της κατανάλωσης οπωροκυπευτικών προς, προς όφελος των μεταποιημένων προϊόντων έχουν σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο για τη γεωργία αλλά και για την υγεία των πολιτών και τις επισητιστικές συνήθειές μας. Κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό είναι το ότι πρέπει να γίνει έλεγχος κατά πόσο προϊόντα τρίτων χωρών να ε, καλύπτουν τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και η παραγωγή της Ένωσης, όχι μόνο φαρμακευτικά και υγειονομικά αλλά και για την ευημερία των ε, ζώων. Τα στοιχεία της ανακοίνωσης Επιτροπής δείχνουν ότι εν ώψη της συνολικής μείωσης της ε, έκτασης των καλλιεργειών για προκυβευτικά υπάρχει και το θέμα της, ε, του μέσου όρου έκτασης αναεκμετάλλευση. που σημαίνει ότι ε, μειώνεται η δυνατότητα, η δύναμη των μικρών παραγωγών σε σχέση με τους μεγάλους. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη οι οργανώσεις παραγωγών θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια καλή λύση αντιμετώπιση του προβλήματο Στον τομέα των αποδοκιβευτικών η κατηγορία αυτή είναι πολύ αδύναμη σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ διαπραγματεύσει. Οι ενώσει παραγωγών ωστόσο πρέπει να γεννηθούν από τα κάτω, να μην συνδέονται με τις ενώσει. Ε, με τις επαγγελματικές οργανώσεις. Οι ενώσει παραγωγών δεν χρειάζεται να, πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να βοηθήσουν στην ε, προσέγγιση και με τους καταναλωτές, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό βοηθά την μείωση της διασπάθησης ε, και, της, ε, και την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι η μεταρρύθμιση του κλάδου έχει να κάνει και με το ζήτημα της επιμελητίας των μεταφορών που πρέπει να το δούμε επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γλέζος, παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν γυρίσετε σήμερα τις αγορές όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποροκυπευτικά προϊόντα, θα δείτε ότι υπάρχουν προϊόντα από όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από την Ευρώπη. Καταγγέλλω ότι εδώ και 30 χρόνια εξακολουθεί μια απαράδεκτη πολιτική εναντίον των, των χωρών του Νότου της Ευρώπης που ενώ παράγουν οπωροκυπευτικά προϊόντα δεν βρίσκονται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθείται η πολιτική που λέει στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην, ε, στο Ισραήλ. Μην αγοράζετε βιομηχανικά προϊόντα από τις Ηνωμένε Πολιτείε και από την Ιαπωνία. Αγοράζετε από εμά και αντί να πληρώνετε με χρήμα δεχόμαστε να παίρνουμε προϊόντα σας. Ως αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης πολιτικής είναι να την πληρώνουν οι παραγωγή αγροτικών προϊόντων της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο σαπίζουν τα προϊόντα στην Ελλάδα τα οποροκυπευτικά και δεν βλέπω αντιμετώπιση από την πλευρά ούτε της, της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του τεράστιου θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας είναι και σκιώδης Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το αξιόλογο έργο του. Άπτεται σημαντικών θεμάτων, το βαθμό οργάνωσης ε, του γεωργικού κλάδου, τις επενδύσεις, την κατανάλωση. Πολύ σημαντικά θέματα. Είναι θετική η εκτίμηση όμως που, στην οποία καταλήγει η έκθεση και αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος γιατί ε, ουσιαστικά λαμβάνει η χώρα μια απελευθέρωση, μια φιλευθεροποίηση της αγοράς εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε με πιο επικριτικό τρόπο αυτή τη διαδικασία απελευθέρωση του κλάδου που δημιούργησε τεράστιες ε, ανισότητες και αδικίες στην κατανομή της παραγωγικής δυνατότητας μεταξύ των περιφερειών και χωρών. Ε, οδήγησε σε στην ανεργία πολλούς γεωργούς που εγκατέλειψαν τη γεωργική δραστηριότητά τους, οδήγησε σε ανεργία στο κλάδο και δημιούργησε μια παράδοξη κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει έλλειμμα γεωργικό, έχουμε μια παραγωγή που μειώνεται σε όγκο, σε αξία και σε επιφάνεια, μειώνεται η κατανάλωση και ταυτόχρονα έχουμε και ενισχύσεις που δεν χρησιμοποιούνται, 4,1% ε, του συνόλου, των, του συνόλου της αξίας, και ουσιαστικά μόνο ένα τρίτο των ε, ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν τελικά στους παραγωγούς. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ε, αδιανόητο και θα πρέπει να το στυλιτεύσουμε. Γιατί έχουμε μέτρα που θα μας επέτρεπαν να επιλύσουμε κάποια προβλήματα. Αλλά όλα αυτά συνδέονται και με τη διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς. Μιλήσαμε για μείωση της κατανάλωσης η κατανάλωση δεν μειώθηκε μόνο εξαιτία της κρίσης. Υπάρχουν και άλλες λόγες. Γιατί σίγουρα μία σούπα λαχανικών δεν είναι πιο ακριβή από ένα χάμπουργκερ. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στα χάμπουργκερ γιατί ε, έξω από τα σχολεία υπάρχουν εστιατόρια οι αλυσίδε fast food που πουλά χάμπουργκερ. Είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση. Μιλήσαμε για τα προβλήματα της αγοράς ουσιαστικά κρατάει χμάλω τους, τους γεωργούς και τους υποχρεώνει σε εγκατάλειψη γεωργικής δραστηριότητας, γιατί γίνονται έρμεα των ε, μεγάλων αλυσίδων διανομής που δεν επιτρέπουν μια ισότιμη κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος ε, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας ανεφοδιασμού των τροφίμων. Επίσης να διαρωτηθούμε γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό οργάνωσης και γιατί έχουμε τόσο κόστος μεγάλο που ε, επιβάλλουμε και κυρίως γραφειοκρατικό στις οργανώσεις παραγωγών και εμποδίζουμε τη μεγαλύτερη οργάνωση, υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, φορολογικά εμπόδια, νοσμολογικά, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια κοινωνικής αναβάθμισης για να αναβαθμίσουμε την οικογενειακή γεωργία, τη γεωργία της μικρής κλίμακος, γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά του παραγωγικού μας συστήματος. Και επίσης πολλές φορές δυστυχώ οι ενισχύσεις δεν φτάνουν σε αυτόν που τις χρειάζεται. Ευχαριστώ. Δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στους και ηγητές, αλλά παρακαλώ μην κάνετε κατάχρηση. Παρακαλώ 1,5 λεπτό στον καθένα. κυρία Πετήρ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Μέλο, τον εισηγητή, για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του. Θεωρώ ότι εντόπισε στην έκθεσή του τα σημαντικότερα προβλήματα του τομέα απορροκυπευτικών ε, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μερικές φορές και γενικώ τον προβληματισμό για τις οργανώσεις παραγωγών. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ε, ώστε να ενθαρρύνουμε και τις ε, κρατικές, τις εθνικές αρχές να απλουστεύσουν τις διαδικασίες. Εμείς στην Κροατία έχουμε μόνο δύο οργανώσεις παραγωγών μία στο γαλακτοκομικό τομέα και άλλη στον απορροκυπευτικό τομέα. Ενώ έχουμε πολλούς γεωργούς που θέλουν να γίνουν μέλη σε οργανώσεις παραγωγών, αλλά εξαιτία της υπερβολικά περίπλοκης διαδικασίας ε, αποτρέπονται, γιατί είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία και τελικά ε, εγκαταλείπουν αυτή τη φιλοδοξία να γίνουν μέλη σε οργανώσεις παραγωγών. Οπότε αυτό το μήνυμα θα πρέπει να στείλουμε προς τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Ε, το αναφέρει στα σημεία 6 και 7 ο κύριος ε, Μέλο, δηλαδή απλούστευση της διαδικασίας και ενισχύσεις στις οργανώσεις παραγωγών για να στηριχθούν και οικονομικά, να οργανωθούν καλύτερα και να είναι πιο ανταγωνιστικές αυτές οι οργανώσεις παραγωγών στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλάιερ. Voorzitter, Op de eerste plaats <clears throat> wil ik graag natuurlijk Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Μέλου. Βεβαίως ε, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις ε, επιπτώσεις της ε, κρίσης με τη Ρωσία. Είναι δύσκολο να υπάρξουν Αποζημιώσεις. Έχουμε πολλά προβλήματα στα οποροκυπευτικά στη χώρα μου, την Ολλανδία. Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, αλλά είναι πολύ δύσκολη η γραφειοκρατία για να μπορέσει να λάβει κανείς αυτές τις αποζημιώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι μηχανισμοί για τη λήψη αποζημιώσεων να απλοποιηθούν. Και για τους οργανώσεις παραγωγών είναι σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα αυτή αυτοοργάνωση ε, η παραγωγή και βεβαίως θα μπορούν να αποφασίσουν και από μόνοι τους οι παραγωγοί πώς θα αξιοποιήσουν τις ε, επιδοτήσεις που λαμβάνουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλο με τον οποίο συμφωνώ για τους, ε, τις βασικές κατευθύνσεις της έκθεσης Συχνά ε, ήδη αναφέρθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει ο χαμηλός ε, βαθμός οργάνωσης του κλάδου που σημαίνει ότι οι πολλοί παραγωγοί δεν έχουν υποστήριξη σήμερα. Οι μικροί παραγωγοί μάλιστα είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο γιατί οι ίδιοι δεν διαθέτουν διαπραγματευτική ε, δυνατότητα ε, στην αλυσίδα παραγωγής. Και είναι εκ των πραγμάτων και η πιο εκτεθειμένη εν ώψη και της παγκοσμιοποίησης. Για να συμπληρώσω το κείμενο θα θέσω τέσσερα στοιχεία για την βελτίωση των τάσεων που περιλαμβάνει ήδη η έκθεση. Πρώτον, να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα των ε, επαγγελματικών οργανώσεων. Να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των εμπορικών αξιών των προϊόντων Αναφέρθηκε γι' αυτό. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη βελτίωσης των εργαλείων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, κάτι ουσιαστικό. Και τέλος, απλοποίηση, απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου στον κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταντάν. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του. Να υπενθυμίσω επίσης ότι με την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, το Κοινοβούλιο και εμείς ιδίως, είχαμε υποβάλει και εγκρίνει μια σειρά προτάσεων που δεν υιοθετήθηκαν ωστόσο εν τέλει στους τριλόγους. Κάποια κράτη είχαν ε, δείξει ότι δεν τους άρεσε ιδιαίτερα ε, το θέμα των οργανώσεων παραγωγών. Η διοικητική περιπλοκότητα σχετίζεται και με την λειτουργία των οργανώσεων σε σχέση με το δίκαιο ανταγωνισμού. Σας τονίζω την ανάγκη την, ε, τη που συνεχίζονται για το δίκαιο ανταγωνισμού και που αποτελούν αντικείμενο της ε, μελλοντική συζήτησης του, της Επιτροπής μας. στο Κοινοβούλιο είχαμε τονίσει ότι μπορεί να υπάρχουν παρεκκλήσεις βάσει τη συνθήκη της Λισαβόνα για να μπορούν να έχουν μια παρέκκληση στο δικαίωμα ανταγωνισμού οι οργανώσει παραγωγών ενώ είναι σημαντικό να λάβει υπόψη επιτροπή και την απόκληση μεταξύ κόστους παραγωγής και φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων που υπάρχουν από χώρα σε χώρα, κάτι που σε κάποια κράτη καθιστούν τις οργανώσεις παραγωγών μη λειτουργικέ. Γιατί οι τιμές παρέμβασης καθορίζονται πολύ υπερβολικά χαμηλά σε σχέση με το κόστος παραγωγής για κάποια προϊόντα. Στο μέλλον πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε για να, υπάρχουν, να υπάρχει κόστος παρέμβασης που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές, τα διάφορα επίπεδα ζωής μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. όταν εγκαταλείπουμε τις δημόσιες πολιτικές και αφήνουμε ανεξέλεγκτη την αγορά, η διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών αποδυναμώνεται και μάλιστα με αλματώδη βήματα. Από αυτή την άποψη, ο οργανώσεις παραγωγών που σχεδίασε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε επινοήσει τότε, ουσιαστικά απλώς συγκαλύπτουν μία πραγματικότητα που κρύβεται καθημερινά οι παραγωγοί, άνδρες και γυναίκες, λαμβάνουν πολύ πιο χαμηλές τιμές ε, για τα προϊόντα τους και έχουν πολύ μικρότερη ικανότητα επιβίωσης. Και στο μέτρο που δεν ε, είμαστε ικανοί να κάνουμε μια κριτική ανάλυση ε, το που οδηγήσαμε τον κλάδο των παραγωγών με τις πολιτικές απελευθέρωσης, αν δεν κάνουμε προηγουμένως αυτή την κριτική ανάλυση δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Και αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε τις τιμές στο επίκεντρο των γεωργικών πολιτικών, τότε θα τα βρούμε πολύ σκούρα. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, αλλά δυστυχώς λείπουν από την έκθεση όλες αυτές οι σκέψεις και όλες αυτές οι κριτικές αναλύσεις και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, δεν θα πρέπει να συνδέσουμε τις ενισχύσεις ε, σε κατάσταση κρίσης, όπως ήταν αυτή με το ρωσικό εμπάργο, ε, από την ε, οργάνωση σε οργανώσει παραγωγό. Θα πρέπει να είναι ελεύθερη απόφαση. Αν ο παραγωγός δεν οργανώνεται σε συνεταιρισμούς οργανώσει, σημαίνει ότι δεν είναι οι οργανώσει ελκυστικέ για αυτόν και ότι δεν του λύνουν τα προβλήματά του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ουαζό. Ευχαριστώ. Η κατάσταση του κλάδου, όπω ξέρετε, παρουσιάζει πολύ μεγάλε διακυμάνσει. Δεν είναι δυνατόν να μας ικανοποιείται ότι μειώνονται οι εκμεταλλεύσεις και οι, οι εκμεταλλεύσεις και οι ε, επιφάνειες. Και άρα δεν μπορούν ούτε καν να καλύψουν οι παραγωγοί στη Γαλλία τις εσωτερικές ανάγκες και κάνουν εισαγωγές. Οι μισές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν καμία δυνατότητα επενδύσεων. Φέτος χρειάστηκε να πουλήσουν τα προϊόντα τους κάτω από την τιμή κόστος η παραγωγή. Κάτι άλλο θα πρέπει να μας ανησυχεί επίσης. Για να καταπολεμήσουμε την πίεση από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι παραγωγοί δημιουργούν τα δικά τους σούπερ μάρκετ που έχουν μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία. Και οι παραγωγοί με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν το διπλό ή το τριπλό από ό,τι θα κέρδιζαν αν πουλάγαν τα προϊόντα τους στα σούπερ μάρκετ και δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα έπρεπε να τις προωθήσει η Κομισιόν. Είναι η απόδειξη ότι η κοινή γεωρική πολιτική σα έχει απορριφθεί από τον κόσμο όπως και το οικονομικό σας σύστημα. Ευχαριστώ κύριος Βαλκάρσελ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους που συνεχάρισαν τον συνάδελφο Μέλου για αυτή τη θαυμάσια εργασία, τη θαυμάσια έκθεση. Οπωσδήποτε ο κλάδος έχει μεγάλη σημασία για πολλές χώρες της Ένωσης, κυρίως ε, χώρες της Μεσογείου. Και στη δική μου, στην περιοχή της Μούρθια στην Ισπανία, παράγονται πολλά οποροκυπευτικά. Είναι πυλώνας και οικονομικός και κοινωνικός, γιατί δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Οπότε, επειδή είναι σημαντικός ο τομέας, οπωσδήποτε πρέπει να εμείνουμε σε ορισμένα θέματα, να ενισχύσουμε τις οργανώσεις των παραγωγών να τους ενισχύσουμε περισσότερο όσον αφορά τις αποσύρσεις ε, παραγωγής, ιδιαίτερα λόγω της ε, μεγάλης ε, διακύμανσης στις τιμές, ούτως ώστε οι πιέσεις αυτές να απαλυνθούν. Οι πιέσεις που υφίστανται από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και άλλοι το ανέφεραν. Προσπαθούν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά έχουμε και τα προβλήματα που δημιούργησε το εμπάργκο για τη Ρωσία. Δεν υπήρξε ικανοποιητική βοήθεια για το θέμα αυτό για τους παραγωγούς μας από την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Εράς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε ένα καλό καθεστώς οπροκυπευτικών σήμερα που μπορούμε να βελτιώσουμε βέβαια. Και μπορούμε να βελτιώσουμε προς την κατεύθυνση που προτείνει ο εισηγητής κ. μέλο. Το κείμενό του είναι πολύ καλό και ευχαριστούμε για την δουλειά που κάνει κύριε Μέλο. Αξίζει η προσπάθεια αυτή. Στην... Σχολιάστε την ανάγκη να αυξηθεί η βοήθεια προς τους οργανώσεις παραγωγών. Συμφωνώ. Και η ιδέα που ακούστηκε να γίνει ανάλυση του, ότι δεν του γιατί δεν χρησιμοποιείται επαρκώς το σύστημα αυτό και πώς μπορεί να βελτιωθεί είναι χρήσιμη. Επίσης, μιλήσατε για την ανάγκη αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες. Να υπάρχει δηλαδή υποχρέωση παραγωγών τρίτων χωρών να τηρούν τι ίδιε προποθέσει με του παραγωγού τη Ένωση. Επίση, συμφωνώ μαζί σα όταν είπατε ότι οι οργανώσει παραγωγών πρέπει να παίξουν ένα ρόλο στην αλυσίδα διατροφή. Είναι ένα μόνιμο θέμα αυτό. Η κυρία Μαγκίνε είναι υπεύθυνη για την σχετική έκθεση. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, αλλά συμφωνώ με κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση τη αλυσίδα διατροφή στην Ένωση. Θα υποβάλουμε τροπολογίε, βέβαια, αυτονόητο, για την αναθεώρηση των τιμών απόσυρση, για παράδειγμα, που πρέπει να επικαιροποιηθούν, την συμπερίληψη τη μεταποίηση σαν ένα ε, από τους στόχους της απόσυρσης και άλλα θέματα, όπως κοινοτικό ποσοστό, χρήση κάποιων κοινοτικών πόρων για την απόσυρση. Σε κάθε περίπτωση συγχανητήρια και να σας αναγγείλω ότι οι τροπολογίες θα είναι λίγες γιατί πραγματικά η έκθεση είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που είπε προηγούμενο, και να ευχαριστήσω θέλω και τον συνάδελφο Μέλο διότι σε μεγάλο βαθμό η οργάνωση αγοράς για τα οπροκυπευτικά λειτουργεί και είναι καλό το σύστημα και βοηθάει τους παραγωγούς. Και σε μια μελέτη την παρουσίαση της οποίας ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, εδώ υπόθηκε ότι δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν ορισμένοι παραγωγοί. Είναι κρίμα αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί στον κλάδο αυτό το ποσοστό οργάνωσης, διότι η παραγωγή αυτή με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πωλήσουν απευθείας τα προϊόντα τους, οπότε χάνουν αν δεν είναι καλά οργανωμένοι. Είναι ενδιαφέρον μόνο για ορισμένους που δεν θέλουν να συμμετέχουν, για ορισμένους που δεν πουλούν απευθείας τα προϊόντα τους. Η κατάσταση όμως των τελευταίων μηνών και οι επιπτώσεις του εμπάργου για τη Ρωσία καταδεικνύουν ότι είναι σημαντική η διαχείριση των κρίσεων. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τις οργανώσεις παραγωγών, ούτω ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Και ιδιαίτερα στον κλάδο αυτό, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να έχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, μια φράση ακόμη επιτρέψτε μου, εάν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, τότε πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ή να αναπτύξουμε άλλα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις οργανώσεις παραγωγών να δημιουργήσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Ο κύριος Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Ε, τον εισηγητή λοιπόν για την εργασία του, λέει ο κύριος Μπούντα, στις ε, νέες χώρες μέλη. Υπάρχουν κάποιες ε, αντιδράσεις ε, έναντι των οργανώσεων παραγωγών, αντιστάσεις θα έλεγα. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τους παραγωγούς ότι μέσω οργανώσεων παραγωγών έχουν περισσότερη δύναμη. Και θα πω κάτι περισσότερο. Δεν πρέπει απλώς να ενθαρρύνουμε τους μικροπαραγωγούς για να μπουν στις ενώσεις. Πρέπει να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, τους δικούς τους χώρους αποθήκευσης. Είναι πολύ σημαντικό για τους ε, μικρούς παραγωγούς να έχουν χώρους αποθήκευσης και χώρους για τη μεταποίηση των προϊόντων τους. Και επίσης θα μπορούσαν να ε, δημιουργήσουν και ε, μαγαζιά μικρά ή μεγάλα που να πολλούν απευθείας τα προϊόντα τους. Έτσι θα μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία έναντι των ε, διακυμάνσεων που παρουσιάζονται στην παγκόσμια αγορά, τα διάφορα εμπάργκο κτλ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπορούν οι ίδιοι οι παραγωγοί να πολλούν λιανικά τα προϊόντα τους. Ο κύριος Μποβέ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και συγχαίρω τον εισηγητή γιατί επισήμανε μερικά πολύ σημαντικά και βασικά θέματα. Επίσης συμφωνώ με τα σχόλια του Μισελ Νταντά γιατί είναι αναγκαίο να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία συζήτησης για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να συμπεριλάβουμε και νέες δυνατότητες ε, οργάνωσης για τους παραγωγούς ε, και ενίσχυσης της διαπραγματευτικής τους ισχύω. Επανέρχομαι στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ε, υπενθυμίζω ότι είχαμε αντιταχθεί στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Μαρόκο για τα απορροκυπευτικά. Δυστυχώς ε, δεν ε, κυριάρχησε η δική μας γνώμη στην Ολομέλη. Η Επιτροπή Γεωργίας πάντως είχε καταψηφίσει τότε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με το Μαρόκο. Για τα ζενιοκτώνα, Είχαμε πει ότι υπήρχε πρόβλημα με αυτό ε, και υπάρχει κατανα... μείωση της κατανάλωσης που οφείλεται στο γεγονός ότι τα προκυπευτικά συγκεντρώνουν κυρίως το μεγαλύτερο βαθμό φυτοφαρμάκων και ζανιοκτώνων στην αλυσίδα διατροφής. Θα πρέπει να μειώσουμε λοιπόν τη χρήση των φυτοφαρμάκων και εκεί να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας μεταξύ άλλων. Ένα άλλο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η στρέβλωση που υπάρχει μεταξύ των μικρών παραγωγών και των μεγάλων βιομηχανικών δομών προεκυπευτικών. Τέτοιες μεγάλες δομές δημιουργούνται με επιχειρήσεις 40-50 εκταρίων σε θερμοκήπια που, που διαταράσσουν, για να μην πω ότι καταστρέφουν την ισορροπία της αγοράς. Και έχουμε και αγροκτήματα όπου, όπου συμπεριλαμβάνονται και φωτοβολταϊκά στις, στα θερμοκήπια, οπότε τα απορροκυπευτικά γίνονται προϊόν των ενεργειακών προϊόντων. Εκεί υπάρχει πρόβλημα λοιπόν στρέβλωσης σε σχέση με τους μικρούς παραγωγούς και περιπλέκει τις ε, σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Οι παραγωγοί μπορούν οι ίδιοι να κάνουν πολλά για να εξασφαλίσουν το ρόλο του στην αλυσίδα διατροφής και για να αντιμετωπίσουν το τομέα του λιανεμπορίου. Χρειάζεται μεγαλύτερη τεχνολογική ανάπτυξη, αναφέρεται σωστά στην έκθεση ότι πρέπει να μειωθεί η διάρκεια της μετακίνησης των οποροκυπευτικών στην αλυσίδα διατροφής. Ξέρουμε ότι η παραγωγή είναι καλύτερο οργανωμένη σε χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή οπωροκυπευτικών. Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Και τα κράτη-μέλη που μπήκαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια νοοτροπία για να σκεφτούν την ανάγκη μια κοινή προσέγγιση. Στη Σλοβενία δεν υπάρχει σχεδόν καμία οργάνωση παρόν. Τα αποκυβευτικά είναι λοιπόν ένα τομέα που μπορεί να δώσει θέση εργασία στο μέλλον. Γιατί έχουμε μικρή σχετικά έκταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νέων θέσεων εργασίας και εγώ προσωπικά θα φέρω κάποιους εκπροσώπους παραγωγών ε, στις Βρυξέλλες και θα τον καλέσω τον κύριο Μέλλον να παρουσιάσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και ο υποφαινόμενος. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ο τομέα των απορροκυπευτικών, για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν είναι ευαλείωτα τα προϊόντα, ευπαθή, και έχουμε και τις πολύ αρνητικές ε, εμπειρίες ε, της περασμένης χώρα, χρονιάς. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο σημαντικοί είναι οι μηχανισμοί διαχείρισης των κρίσεων. Και χρειαζόμαστε και παρέμβαση στην αγορά. Είναι σημαντικό το θέμα και της παρέμβασης ε, στα πλαίσια της διαχείρισης των κρίσεων. Επίσης, να ενισχύσουμε την κατανάλωση των απορροκυπευτικών, που έχει μειωθεί. Και επίσης, για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα πρέπει να εισαγάγουμε και νέους μηχανισμούς. Επίσης, ε, τα μηδέα κεφάλαια είναι ένας ε, τρόπος ε, ή κάποια χρηματοοικονομική ενίσχυση για να αποκατασταθεί αυτή η σταθερότητα. Επίσης, θα πρέπει να στηρίξουμε συγκεκριμένα και τις οργανώσεις παραγωγών. Όλες αυτές οι ενέργειες πιστεύω ότι θα αποφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κορτέ, τον Διευθυντή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου Μέλου και η Επιτροπή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις ε, συστάσεις του και κυρίως με την έκκληση που κάνει για περαιτέρω ενδυνάμωση των οργανώσεων παραγωγών, ούτω ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να είναι και πιο ελκυστικές οι ενώσεις για τους παραγωγούς και επίσης να είναι πιο ελκυστική η δημιουργία τέτοιων ενώσεων. Σε ένα βαθμό έχουμε επιτύχει. Αν δείτε τα στοιχεία που τα αναφέρει και η έκθεση μέλου, ο βαθμός οργάνωσης αυξήθηκε από 31% το 2007 σε 43% το 2010 και το 2012 φτάσαμε το 47%. Άρα λειτουργεί η πολιτική μας σε ένα βαθμό. Αλλά υπάρχουν τρομερές ε, ανισότητες όπως βλέπουμε από τους πίνακες μεταξύ κρατών μελών. Και γενικά, σαφώς, 47% είναι ακόμη ανεπαρκές. Και το ρωσικό εμπάργο, όπως πολλοί βουλευτές είπαν σήμερα το πρωί, κατέστησε απόλυτα σαφές ότι η ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών στον κλάδο είναι πολύ σημαντική. Διότι ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε οποιασδήποτε μεταβολές στην αγορά τα προϊόντα είναι ευπαθή και πολλούνται απευθείας στους λιανοπολιτές. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης. Γι' αυτό υπάρχει τεράστια ανάγκη να ενισχύσουμε τη θέση των παραγωγών δύο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, η έκκληση για περαιτέρω απλούστευση κατά πολέμηση λοιπόν της γραφειοκρατίας. Και δεύτερον θα πω και μερικά λόγια για θέμητες εμπορικές πρακτικές. Για το πρώτο. Είναι σαφές. Και καλωσορίζω αυτά που λέει ο κύριος Μέλλον στην έκθεσή του γι' αυτό. Είναι σαφές ότι ο Επίτροπος και γενικά η Επιτροπή στοχεύουν στην περαιτέρω απλούστευση της κοινή οργάνωσης αγοράς, γενικά των κοινών οργανώσεων αγορών συμπεριλαμβανομένων και των οπορικευτικών. Ο κύριο Χόγκαν συντόμω θα σα αποστείλει και εσά και στο Συμβούλιο μια επιστολή που θα παρουσιάζει πολύ πιο αναλυτικά τι απόψει του επ' αυτού. Τι θα κάνουμε. Σε έναν βαθμό ήδη το κάνουμε φέτο. Είναι μια αρκετά εκτεταμένη απλούστευση στα οπορκευτικά για την ε, νομοθεσία που εγκρίνει η ίδια η Κομισιόν, δηλαδή την δευτερογενή τους εφαρμοστικού κανονισμού δηλαδή και τη κατεξοδότηση πράξη. δηλαδή. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιοδό. προς την κατεύθυνση ακριβώς ε, που προτείνει ο κύριος Χάιτεμα και άλλοι. Αλλά, αλλά, πρέπει να είμαι ειλικρινή. τα πιο σημαντικά περιθώρια πλούστευση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Άρα πρέπει να δούμε και τις ε, πρωτογενείς πράξεις, το πρωτογενές δίκαιο που φυσικά υποβάλλονται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο Επίτροπος, όπως είπα, ε, ιδιαίτερος προσεχώς θα σας παρουσιάσει τις ε, ιδέες όσον αφορά την τροποποίηση του βασικού νόμου, ιδιαίτερα το επίπεδο στήριξης των οργανώσεων παραγωγών και για τις αποσύρσεις σε περιπτώσεις κρίσης. Σε τι βαθμό μπορεί να αντισταθμίσει ο ενωσιακός προπολογισμός. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στη βασική νομοθεσία, στο βασικό νομοθέτημα. Άρα δεν μπορεί να το κάνει μόνη της Επιτροπή αυτό το έργο απλούστευσης. Τώρα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που αναφέρθηκαν από πολλούς από τους ε, αξιότιμους βουλευτές σήμερα το πρωί, συμφωνώ με αυτά τα σχόλια και επιβεβαιώνω ότι ο Επίτροπος Χόγκαν θέλει οπωσδήποτε να κάνει. Είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά και η έκθεση της κυρίας Μαγκίνες θα είναι πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε. Να ενισχύσουμε το ρόλο των παραγωγών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Σε σχέση με το λιανεμπόριο. Έχουμε ήδη την πρωτοβουλία για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Και ε, μέχρι τέλους του χρόνου η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορα περαιτέρω βήματα. Να δούμε καταρχάς τι έχει ήδη συμβεί σε αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού και να δούμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Επίτροπο Χόγκαν, διότι ξέρετε, τρόφιμα δεν είναι μόνο θέματα γεωργίας, αφορούν και αρμοδιότητες άλλων επιτρόπων. Ευχαριστώ πολύ. Και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συζήτησης αυτού του σημαντικού θέματος με τον κύριο Μέλου και την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο μετά το σχόλιο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επισημάνω ότι δίνουμε μάχη στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γεωργίας για να διεκδικήσουμε καθήλια αρμοδιότητα από κοινού με την ε, Επιτροπή Ιστορικής ε, Αγοράς με βάση το άρθρο 54 και ξέρω ότι το προωθεί ο Πρόεδρος γιατί αν δεν κερδίσουμε τώρα αυτόν τον αγώνα, αυτή τη μάχη ο ρόλος της ε, Επιτροπής μας στο μέλλον θα είναι πολύ αποδυναμωμένο σε σχέση με την αλυσίδα εφοδιασμού και θα πρέπει ο γεωργικό Κλάδο να αναγνωριστεί ως βασικό σημείο αφετηρίας της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα και υπάρχουν δυστυχώ πολλοί ευρωβουλευτέ που διαφωνούν. Και ακόμη και στην ε, Επιτροπή υπάρχουν ε, άνθρωποι που δεν είναι αυτή τη γνώμη. Θα έλεγα λοιπόν να δώσουμε από κοινού τη μάχη, στηρίζοντα τον πρόεδρό μα, προκειμένου να αναγνωριστεί η θέση μα στη συζήτηση αυτή. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η μάχη, θα πρέπει να τη δώσουμε τώρα, γιατί αν τη χάσουμε τώρα θα μείνουμε πολύ πίσω. Και ευχαριστώ που ε, αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να ζητήσω την αμέριστη και συνεχή υποστήριξή σας στη μάχη μας. Ναι, το συζήτησα με τον ε, πρόεδρο Μπούζεκ και θα εμπλουτίσουμε την επιχειρηματολογία μας παίρνοντας το θέμα στην Επιτροπή, ε, στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Όπως σας είπα το έθεσα στον Πρόεδρο Μπούζεκ. Ε, δεν ξέρω Κύριε Νούνο, δεν έχετε πια χρόνο, γιατί λάβατε τέτοια εγκόμια και πένους που εξαντλήθηκε ο χρόνος που είχαμε για το σημείο αυτό στη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο σύντομα, παρακαλώ. Θα είμαι πολύ λακωνικός. Σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τα σχόλιά σας. Ήμουν πριν επιγραμματικός, το ίδιο θα κάνω και στα συμπεράσματα. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη της έκθεσης. Ε, σημείωσα 19 ομιλητές, 19 παρεμβάσεις, δεν είναι και λίγο. Και ε, συζήτησα το θέμα αυτό με τους και και κατάγραψα με λεπτομέρειες τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα και πραγματεύεται πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και πολλές πτυχές. Εγώ συγκράτησα τέσσερα-πέντε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους ευρωβουλευτές. Για παράδειγμα, η διαχείριση των κρίσεων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το σχέδιο έκθεσης και στην αιτιολογική έκθεση και στο διατακτικό μιλάει με σαφήνεια για την ανάγκη διαχείρισης της κρίσης. Αναφέρθηκε και η κρίση με τη Ρωσία. Και μάλιστα αναφέρεται ότι το ρωσικό εμπάργο άσκησε αρνητικές συνέπειες στον απορροκυρευτικό τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται μία ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών ώστε να, να μπορέσουν συλλογικά να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες ε, και απροσδόκητες καταστάσεις. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι τα μέσα διαχείρισης κρίσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των ευρωπαϊκών, δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Και έχουμε δύο συγκεκριμένες αιτιολογικές σκέψεις, την 12 και τη 13 που αναφέρονται στη διαχείριση των, της κρίσεως, των κρίσεων. Συγγνώμη. Θα πρέπει να ε, δικαιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν χρησιμοποιεί επαρκώ ε, τα μέσα διαχείριση κρίσεων και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστε πρακτικέ ε, των εφισταμένων οργανώσεων παραγωγών. Επίση, να συμβάλλει σε επιλέξιμα αμοιβαία κεφάλαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί καλύτερα τι κρίσει και να προστατεύσει καλύτερα του παραγωγού σε περίπτωση κρίση ιδιαίτερα σε κρίσεις που αποδυναμώνουν τα γεωργικά εισοδήματα. Και αναφέρθηκε το θέμα του γεωργικού εισοδήματος ε, και του εισοδήματος των παραγωγών. Αυτό θα το προωθήσουμε και μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Αυτό το αναφέρω στην ε, έκθεση και μέσω της διαχείρισης των κρίσεων, αλλά και μέσω των σχέσεων των παραγωγών με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και από αυτή την άποψη σας παραπέμπω στο σημείο 2. Ε, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να καταπολεμήσει αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα διανομής τροφίμων που έχουν αρνητική συνέπεια στο γεωργικό εισόδημα, μειώνει τους μισθούς και αποδυναμώνει τη δυνατότητα επιβίωσης του τομέα. Φαίνεται λοιπόν στην έκθεση ότι έχει νόημα η οργάνωση σε οργανώσεις παραγωγών και βοηθά στην ε, αύξηση του γεωργικού εισοδήματος μια τέτοια οργάνωση. Δεν πρόκειται να επεκταθώ τώρα περαιτέρω, ούτε θα ασχοληθώ με ιδεολογικά ζητήματα. Γιατί κάποιοι αφισβήτησαν την απελευθέρωση του κλάδου. Αυτό το ζήτημα είναι ιδεολογική υφή. Αυτό που εξετάζει η έκθεση είναι το θέμα των οργανώσεων παραγωγών. Δεν μπορώ να μετατρέψω μια έκθεση για τις οργανώσεις παραγωγών που έχει ως πρωταρχικό στόχο την, την ε, παρότριση των παραγών να οργανωθούν για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, αυτή την έκθεση να τη μετατρέψω σε κάτι α, ε, τελείως διαφορετικό, που ουσιαστικά την αλλοιώνει και για να πω ότι την εξουδετερώνει κιόλα. Ξέρω ότι υπάρχουν χρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οργανώσεις παραγωγών. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για να ενισχυθούν. Και δεν θα πρέπει να παρατερίνονται και να εξωθούνται στην απομόνωση η παραγωγή. Η έκθεση μου, επαναλαμβάνω, αφορά τι οργανώσει παραγωγών και σε αυτό το θέμα θα επικεντρωθώ. Θέλω να ε, συνεχίσουν να λειτουργούν και να βελτιωθεί η λειτουργία του στο μέλλον. Και αν υπάρχουν δυσλειτουργίε, αυτέ να διορθωθούν. Τώρα, αν κάποια στιγμή έχουμε άλλη έκθεση με θέμα την απελευθέρωση του κλάδου, τότε να μιλήσουμε για την απελευθέρωση. Αλλά άλλο είναι το θέμα τη δική μου έκθεση. Είναι οι οργανώσει παραγωγών και σε αυτό θα περιοριστώ. Επίση, ε, και το θέμα τη ανανέωση τη γεωργίας είναι πολύ εύστοχο, αλλά δεν είναι αντικείμενο τη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν μπορεί να μιλά αυτή η έκθεση επί παντός Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη το θέμα της γύρασης και να ενισχύσουμε τους νέους. Έναν ε, νέο μόνο Γεωργό έχουμε στην, ε, στην Γεωργία για εννέα που αποχωρούν. Αλλά είπαμε, δεν είναι αυτό το αντικείμενο της έκθεσης. Εμείς ασχολούμαστε εδώ με τις οργανώσεις παραγωγών και θεωρούμε ότι αυτές είναι ευκαιρία για τη βελτίωση και του μέλλοντος της γεωργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους για τους επένους τους, γιατί πραγματικά με ενθαρρύνουν και με ψυχώνουν για να συνεχίσω το έργο μου. Και θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας και περιμένω τις προτάσεις σας. Γιατί η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο δικιά μου, είναι η έκθεση ολόκληρη τη Επιτροπή Γεωργία ε, και στόχο μα είναι να βοηθήσουμε ένα πολύ σημαντικό τομέα όπω είναι τα ποροκυπευτικά. Σα ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να, επαναλάβω κάτι, να κάτι που είπε ο κύριος Μποβέ. Στον τομέα αυτών των ποροκυπευτικών κυριαρχούν οι μικροί παραγωγοί. Γι' αυτό και χρήζουν ιδιαίτερη υποστήριξη αυτή η μικρή παραγωγή και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την οργάνωσή τους σε οργανώσεις παραγωγών το είναι πολύ σημαντική αρχή και απαιτεί διαφορετικό επίπεδο στήριξης. Θα ήθελα λοιπόν και ο εισηγητής και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δουν αν υπάρχουν και εναλλακτικέ ε, ε, μέθοδοι στήριξη των μικρών αυτών παραγωγών που επαναλαμβάνω κυριαρχούν στο τοπίο των απορροκυπευτικών. Ευχαριστώ. Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι έχετε προθεσμία για να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις ε, της ε, διατλαντικής εταιρικής σχέσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις. τη TIP τα αρχικά. Στην τελευταία μας συνεδρίαση τον Ιανουάριο διοργανώσαμε μία ανταλλαγή απόψεων επί της ε, γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Γεωργίας ε, στην ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, που είναι η αρμόδια καθήλη για το θέμα αυτό. Η έκθεση της ΣΥΝΤΑ θα περιλαμβάνει κάποιες στάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις της πολύ σημαντικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης του TTIP για το εμπόριο και τις, τις που θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Τεράστιες προκλήσεις, εξαιρετικά σημαντικό το θέμα, γι' αυτό και μερικοί περιμένουν ε, η οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταφερθεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει φυσικά στο πλαίσιο αυτό να εξεταστούν τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας και να ληφθούν υπόψη οι απειλές προς τον γεωργικό τομέα από ενδεχόμενη συγκεκριμένη τροπή της συμφωνίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συγκητές μας για να μας ενημερώσουν για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό, όπως σας είπα, θέμα και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Δεν ξέρω ποιο θα λάβει πρώτο το λόγο. Ο κύριο Δεκάστρο ή ο κύριο Νίκολσον. Κύριε Δεκάστρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η άποψη, η σύσταση που παρουσιάσαμε τον κύριο Νίκολσον είναι μία σελίδα. Γι' αυτό θα προσπαθήσω μαζί με τον Τζιμ σε λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω τη δουλειά που κάνουμε. Κάτι που δεν είναι εύκολο, ιδίως μετά τη συζήτηση που είχαμε τη στην περασμένη συνάντηση της Επιτροπής μας. Ξεκινήσαμε το κείμενο με τρεις αιτιολογικές σκέψεις που πρέπει να είναι η βάση πάνω στην οποία θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις στην Επιτροπή Ίντα για αυτό το λεπτό και σημαντικό θέμα των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζουμε καταρχά ότι ο κλάδο τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ουσιαστικό και εξαιρετικά λεπτό τμήμα των ε, διατλαντικών διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Θυμίζουμε ότι καταγράφονται ε, σημαντικές εμπορικές ε, πλεονάσμα με τη ΣΥΠΑ και από τις διαπραγματεύσεις αυτές μπορεί να κερδίσει η ευρωπαϊκή γεωργία με μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην αμερικανική αγορά. Το δεύτερο σημείο αφορά την ε, ανάγκη, την απόλυτη ανάγκη που υπογραμμίζουμε στη νομοδότησή μας να μην αλλάξουν να μην αλλάξει σε κανένα σημείο τα επίπεδα ποιότητας που έχουμε στην Ευρώπη που αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινώντας από την αρχή της προφύλαξης. Και δεν πρέπει να τεθούν σε αμφισβήτηση, ούτε θέλουμε να τεθούν σε αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της, ε, των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αφετέρου, υπάρχουν πολλά, όχι μόνο δασμολογικά, αλλά και υγειονομικά εμπόδια που εμποδίζουν τις ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διαπραγμάτευση αυτή πρέπει να είναι θετική και για τις δύο πλευρές και να επιτρέψει να μειωθούν τα φυτοϊγειονομικά εμπόδια επιτρέποντας τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κερδίσουν πραγματικά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα υπογραμμίζουμε το ζήτημα των ευαίσθητων προϊόντων όπου θα υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός που θα εξέφεται τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε υπερβολικές πιέσεις ιδίως για κάποια προϊόντα που θα αντιμετώπιζαν προβλήματα από, τη μία, από την αγορά, από το ελεύθερο εμπόριο με τη ΣΥΠΑ, όταν η διαφορά κόστους παραγωγής είναι υπερβολικά υψηλές. Ένα βασικό στοιχείο της γνωμοδότησή μας είναι και το θέμα της ε, σημαντικής αύξησης των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω δε των καλύτερων πληροφοριών και τη καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε να προωθούνται στο εμπόριο στις ΗΠΑ ευρωπαϊκά προϊόντα μπερδεύοντα τους Αμερικανούς ε, παραγωγού λέγοντα ότι είναι ευρωπαϊκά προϊόντα ενώ στην πραγματικότητα είναι αμερικανικά. Άρα το γενικότερο θέμα τη γεωγραφική ένδειξη. Η μνήμα μάλιστα στην πρόσφατη συμφωνία με τον Καναδά στο θέμα αυτό θα ήταν χρήσιμο. Και τέλο, υπογραμμίζουμε το θέμα τη διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρξει πλήρη, ε, ολοκληρωμένη διαφάνεια στι γνώσει των διαπραγματεύσεων, τόσο ώστε το Κοινοβούλιο ε, και εμείς αλλά και η Επιτροπή Ίντα κατόπιν να ξέρουμε τι γίνεται, να κληθούμε, να λάβουμε θέση για το έργο των διαπραγματευτών. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο Πάολο, η γνωμοδότηση αυτή αναφέρει σαφώς τη θέση μας και λέει ότι ο γεωργικός τομέας είναι πολύ ευαίσθητο τμήμα των διαπραγματεύσεων γιατί οι γεωργοί θα ωφεληθούν πολύ αν υπάρξει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση. Οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα πρέπει, πρέπει να γίνει σε βάρος των προδιαγραφών μας για την ασφάλεια των τροφίμων και την ε, ευημερία των ζώων. Ευημερία και ασφάλεια των ζώων. Οι προδιαγραφές μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά παρανοήσεις για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ακούμε για τις ορμόνες, τους ε, τροποποιημένους οργανισμούς, ε, τις χλωριωμένες ε, κότες, αλλά έχουμε και εμείς ε, συμφέροντα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να επιτύχουμε υψηλότερη πρόσβαση για τα υψηλού επίπεδου υψηλού ποιοτικά επίπεδου προϊόντα μας παρά τις αντιδράσεις στην Αμερική θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση λοιπόν για τα υψηλού επίπεδου προστατευόμενα προϊόντα μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδος 3,4 δις. Είναι σαφές από την γνωμοδότηση ότι αυτή είναι μια καλή βάση και είναι πολύ καλό προηγούμενο άριστο η συμφωνία με τον Καναδά. Γιατί στη συμφωνία με τον Καναδά έχουμε συμπεριλάβει 145 προϊόντα υψηλής ε, ποιότητας. Βεβαίως, μπορεί να υποστούμε υπερβολικές πιέσεις από τα αντίστοιχα προϊόντα των ΗΠΑ να υπάρξουν αυτές τις συμφωνίες. Οπότε πρόκειται από πλευρά μου να επερασπιστώ του τομεί αυτούς γιατί δεν νομίζω ότι είναι προς το βράχι μέσο ή πρόθεσμο συμφέρον μας να καταργηθούν τομεί της γεωργίας μας. Οι κύριοι αντίπαλοι μας τα κύρια προβλήματα, κυρίως τα φύτο και, υγειονο... και τα υγειονομικά και φυτο μέτρα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Οι γεωργοί μας οπωσδήποτε αξίζουν μια καλύτερη συμφωνία και εγώ θεωρώ ότι μια ε, δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. νομίζω ότι μπορούμε με πολύ σύντομο τρόπο να επισημάνουμε τα πιο ευαίσθητα ζητήματα και να μείνουμε σε κάποια γενικά θέματα, γιατί ταυτόχρονα ασχολούνται με το θέμα αυτό τέσσερις επιτροπές. Δύο τώρα και δύο θα ασχοληθούν το απόγευμα. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα λοιπόν και ασχολούνται με αυτό πολλές και διάφορες επιτροπές ε, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γιάρ, μετά στην κυρία Σένρα και μετά στον κύριο Σκόν. Ο κύριος Γιάρ. Äh, äh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους Δεκάστρο και Νίκολσον. Και χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει θετική κατεύθυνση γιατί έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε επί των θεμάτων της ουσίας, γιατί μέχρι στιγμή η συζήτηση για το TTIP έχει γίνει μέσω των, μέσων, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν βοηθάει. Γιατί πολλές φορές η συζήτηση στα μέσα δεν ασχολείται με τα ουσιώδη θέματα. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν θέλω λοιπόν να αποτύχουν αυτές οι συζητήσεις λόγω της γεωργίας. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες. Αλλά καθορίζουμε σαφώς και έχουμε συνέστηση και των κινδύνων. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει διαφάνεια στην πληροφόρηση του καταναλωτή. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το βασικό είναι να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει και από πού προέρχεται. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια και για τις δύο πλευρές και αυτό σημαντικό και γι' αυτό με εκνευρίζει στη συζήτηση που γίνεται μέσω του τύπου ότι δεν αναφέρονται ότι ακόμη υπάρχουν εμπόδια στην, στο εμπόριο διότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι γιατί χρειαζόμαστε περαιτέρω συμφωνία όλα λειτουργούν μια χαρά όχι δεν αναφέρεται ότι υπάρχουν εμπόδια που δημιουργούν δυσχέλειες. Τρίτο. Θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση όταν αρχίζουμε να διαπραγματευόμεθα. Οι περισσότεροι έχουμε πάει στις ΗΠΑ. Βλέπουμε πώς γίνονται τα πράγματα εκεί. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε από πλευρά ανταγωνιστικότητα στην Αμερικανική Γεωργία. Είμαστε ισότιμοι συνομιλητές και με αυτή τη βάση πρέπει να διαμορφώσουμε τι διαπραγματεύσει. Κυρίω βέβαια θέλω να πω στον συγκητή μα ενδιαφέρουν τα ευαίσθητα προϊόντα. Ευαίσθητο ήδη εξετάζει, εξηγεί τι είναι. Δεν είναι δυνατόν όμω να θεωρήσουμε ότι όλα τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Γεωργίας είναι ευαίσθητα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ μας τι ακριβώς είναι ευαίσθητο προϊόν. Σε αυτά πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ευχαριστώ η κυρία Σένερα που είναι σκιώδη συγγήτρια. 1,5 λεπτό λοιπόν, η υπόλοιπη από ένα λεπτό. Ε, gracias, ε... Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες πιστεύω σε αυτό το σχέδιο συστάσεων. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος για το TTIP. Δεν ξέρω αν υπήρξε καμία νέα έκθεση, αλλά εδώ στην Επιτροπή μας ακούσαμε μία έκθεση εμπειρογνωμόνων που έλεγε ότι η Γεωργία θα είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της συμφωνίας. Υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος τώρα να θεωρήσουμε ότι θα είναι θετικό το TTIP για τη Γεωργία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Γεωργία είναι πάνω απ' όλα η παραγωγή. Γιατί πολλές φορές ε, τους ξεχνάμε εντελώς τις συζητήσεις μας. Και με ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με ενδιαφέρουν και οι καταναλωτές. Γιατί στο τέλος αυτοί θα πρέπει να αγοράσουν τα προϊόντα. Και νομίζω ότι θα ήταν μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για να δημιουργήσουμε πλούτο για να επιβιώσει αυτός ο κλάδος, να επιβιώσει ύπεθρος. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιχειρούμε να παρουσιάσουμε ως ε, πολύ θετικό, να υποβάλουμε τους γεωργούς μας σε μια σειρά από προδιαγραφές και σε πλήρη επισφάλεια. Διότι εάν συμβούν όλα αυτά όπως ξέρετε και όπως λέει και το ε, παρατηρητήριο για τα γαλακτοκομικά, δεν έχουμε κανένα πλεονέκτημα από μια τέτοια συμφωνία και δεν θα μπορούμε να πουλήσουμε σε κανέναν, ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές χιλιάδες ε, μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις θα εξαφανιστούν. Και επειδή υπάρχει και κλιματική κρίση και μείωση της τιμής του πετρελαίου, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε προϊόντα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Δεν είναι δυνατόν να υποχρέσουμε τους ε, πολίτες μας να τρώνε ζανιοκτόνα και κλωνοποιημένα προϊόντα και τροποποιημένους οργανισμούς και χλωρινωμένες κότες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για λεπτό η τελευταία μας ε, Σκιώδη κυρία Σκότκα. Ευχαριστώ. Ανησυχώ από τον πολύ επιφανειακό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η έκθεση τη γεωργίας με τη μονοσέλιδη έκθεση από ό,τι αφορά τις, από τι γεωργικές ενδείξεις μέχρι τα χημικά. Κατά διάρκεια των ετών, οι πολιτικοί τη Ένωση έχουν διατηρήσει υψηλά επίπεδα στη γεωργία για να επικαλούνται το ότι κάνουμε το καλύτερο τρόφιμα στον κόσμο που είναι καλύτερα, όπως προκύπτει από αυτά που παρέχονται σε την άλλη πλευρά του, του Ατλαντικού. Οι μυστικές διαπραγματεύσεις, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι έτοιμες να θυσιάσουν τα πρότυπα αυτά. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την προσέγγιση αυτή και θα υποβάλουμε τροπολογίες για την προστασία των υψηλών επιπέδων προστασίας των τροφίμων. Μια βασική προϋπόθεση διατήρησης των προτύπων είναι οι διαμετρικά αντίθετοι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουμε το θέμα του κινδύνου πολλοί από τους κινδύνους είναι βασικοί για την δουλειά στη γεωργία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εισαγωγή νέων προϊόντων προϋποθέτει την απόδειξη της ασφάλειας. Αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ακολουθούμε την αρχή της προφύλαξης. Αντίθετα, η Αμερικανική νομοθεσία θεωρεί ότι αν δεν αποδειχθεί η βλάβη, είναι ασφαλές ένα προϊόν. Εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την αρχή της προφύλαξης, που είναι ουσιώδου σημασία για τη διατήρηση του επίπεδου της υγείας και να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ε, υγείας στους ανθρώπους και τα ζώα. Καταγράφουμε ότι ε, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα περνούν αυστηρό έλεγχο στη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην αγορά των ΗΠΑ αυτό δεν συμβαίνει. Ε, φυστούμε την προσοχή σας ότι τα τελευταία έτη η υπηρεσία των τροφίμων της Ένωσης έχει υποβάλει επιφυλάξεις το 30 με το 60% των περιπτώσεων που εξέτασε η βάση του κόντεξ αλιμεντάριους, υπογραμμίζοντας τον υψηλό βαθμό διαφωνίας με τον φυστάμενο με τα στάντα του κώδικα. Γιατί σε προηγούμενες, σε προηγούμενες συζητήσεις, πρόεδρε, οι ομιλητές είχαν τρία λεπτά, εγώ είμαι σκιώδης και δεν έχω τρία λεπτά. Μπορείτε να μου το πείτε γιατί οι πολίτες ανησυχούν για το θέμα της μυστικότητας. Εγώ θα έπρεπε να έχω ένα ακόμα λεπτό για λόγους διαφάνειας. Συνεχίστε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν θα καλύψω από, για λόγους ευγένειας. Πάντως τα θέματα που αφορούν την ε, νομοθετική συνεργασία είναι θέματα στα οποία θα υποβάλουμε τροπολογίες για την προστασία των ε, στάνταρτ. Επίσης, στην ευημερία των ζώων υπάρχει μια σειρά ρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτουν πολλά είδη ζώων σε κάθε φάση της κτηνοτροφίας που δεν υπάρχουν στη ΣΥΠΑ. Ιδίως την υγεία των ζώων αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Συμπερασματικά, Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφου ότι ο ρόλος μας είναι να προστατεύσουμε τα υψηλά επίπεδα γεωργία ό,τι αφορά την ασφάλεια τη υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Η, τα πρότυπα αυτά είναι σε κίνδυνο λόγω της διαδικασία εναρμόνιση με τα πρότυπα στη ΣΥΠΑ ε, με τα οποία μέχρι τώρα οι συγκρίσει ήταν καλύτερες για μας. Εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την ε, ασφάλεια, στην υγεία και στα τρόφιμα. Καλωσορίζω αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί για την υποστήριξη των προτύπων της Γεωργίας της Ένωσης. Θα δούμε κατά πόσον οι θέσεις αυτές θα, γίνουν, ε, θα υλοποιηθούν και στις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Δώσαμε κάποια προτίμηση και προτεραιότητα στους και ηγητές. Τώρα, οι υπόλοιποι από ένα λεπτό. Και δεν χρειάζεται να παραλαμβάνετε αυτά που ήδη ακούσαμε. Ο κύριος Νέκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάου Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τις συστάσεις του κυρίων Ντεκάστρο και Νίκολσον. Η εταιρική αυτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζεται στο νεοφιλελεύθερο δόγμα και αγνοεί τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κάποια χρηματοοικονομικά μέσα για να προωθεί τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείε, Τονίζοντας και ε, ξέροντας την ποιότητα αυτών των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε με γεωργικές εκθέσεις ε, και διαφημιστικές εκστρατείες να προβάλλουμε τέτοια προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τις νέες χώρες ε, που πρόσφατα προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Βουλγαρία, η πατρίδα μου. Οι βούλγαροι παραγωγοί ανησυχούν ιδιαίτερα για τον ε, ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο από τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς αλλά και από τους Αμερικανούς. Ευχαριστώ. Ε, επειδή υπάρχει μια τάση για υπέρβαση του χρόνου αγορεύση, θα σας ε, επαναφέρω στην τάξη με το σφυράκι μου. Κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμμερίζομαι την άποψη των κυρίων Ντεκάστρο και Νίκολσον ότι είναι τόσο θετική η κατάσταση όπως την παρουσιάσατε. Ξέρουμε τη μελέτη του Ινστιτούτου Ιντεφό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου εξετάστηκαν όλες οι επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα. Το TTIP πρέπει να διαμορφωθεί έτσι, ούτως ώστε να μην έχουμε τις χειρότερες επιπτώσεις. Βεβαίως ε, πρέπει να αποφύγουμε την ευθυγράμμιση στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτό θα είχε ως συνέπεια οι οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία να ε, υποστούν μεγαλύτερη πίεση ανταγωνισμού και θα είναι οι χαμένοι. Για τη συζήτηση επί της ουσίας, ε, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Γιάρ, βεβαίως να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αν υπάρχει διαφάνεια. Εφόσον έχουμε διαδίκτυο και κοινωνική δικτύωση, πρέπει οπωσδήποτε οι πολίτες να ενημερώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σμποβέ mm διάβασα με προσοχή το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτο στοιχείο είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι η Επιτροπή Γεωργίας δίνει μόνο γνωμοδότηση στην, εμπορική, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι θλιβερό μόνο γνωμοδότηση. Ο, η σημασία της γεωργίας ξεπερνάει την απλή γνωμοδότηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, έγινε λόγος για τη μελέτη αντικτύπου. Ήταν καταστροφική και επ' αυτού πρέπει να σταθούμε καταστροφική και για τις τιμές και την αγορά και για τα εισοδήματα των γεωργών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τρίτο θέμα. Για μια ακόμα φορά η γεωργία θα αποτελέσει το αντίτιμο για τις υπηρεσίες. Εγώ ζητώ σήμερα ε, σαφώς να απορρίψουμε το TTIP. Μία μόνο είναι η τροπολογία που, που αξίζει. Απορρίπτουμε τη συμφωνία, δεν συμβάλλει τίποτα και καθόλου στην γεωργία και τους Ευρωπαίους γεωργούς. Κύριε Μποβέ, γνωμοδότηση μόνο μία εννοείται. Μπορεί να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, αλλά μόνο μία γνωμοδότηση θα δώσει η Επιτροπή μας εννοείται. Ο κύριος Γλέζος, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο έχω καταγγείλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του εμπορικού ΝΑΤΟ. Η Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Κλίντον έτσι το είχε ονομάσει την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν κατάλαβε το λάθος της έκανε υποχώρηση και έδωσε άλλη ονομασία τη TTIP. Η ουσία είναι ότι εφόσον έχει υπογράψει οι Ηνωμένες με κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδική συμφωνία και εμπορική και για τα αγροτικά προϊόντα για ποιο λόγο χρειάζεται παραπάνω και επιπλέον αυτού του είδους συμφωνία ο μόνος λόγος είναι όπως με το ΝΑΤΟ προσπαθεί να κανοναρχεί και να διοικεί την Ευρώπη το ίδιο προσπαθεί να κανοναρχεί και την, τα εμπορικά της προβλήματα και την εμπορική της διείσδυση στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν προϊόντα, το κατήγγυλα και προηγουμένως, γύρω από την από τα οποροκυπευτικά από, και από τις Ηνωμένε Πολιτείε και σαπίζουν τα οποροκυπευτικά και δεν είδα καμία απάντηση. Δεν πειράζει. Φωνή βόντος εν τη Θα, κάποτε ο λόγος ο σωστός θα βρει το δίκιο του. Ευχαριστώ äh, Ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό που λέει στο τέλος, ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα άλλη μια φορά, αλλά δεν μπορούμε ως βουλευτές να συμμετάσχουμε στην συζήτηση και θα τεθούμε πρώτα τελεσμένων. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Δεύτερον, δεν ε, συζητάμε το ρόλο των μηχανισμών ε, επίλυσης διαφορών. Και δεν αναφέρεται ο κίνδυνος αυτός της ε, συνεργασίας για τα θέματα τα αριθμιστικά. Είναι επικίνδυνα τα θέματα αυτά. Δεν αναφέρονται στην έκθεση. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί που θεωρούν ότι θα έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα έχουν να κερδίσουν και θα διατηρήσουμε τις προδιαγραφές μας, Όλοι όσοι θεωρούν αυτά ε, ότι ισχύουν θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν ισχύει αυτό και ότι αν δεν τους πούμε ότι στους ε, καταναλωτές και τους παραγωγούς μας ότι θα μειωθούν οι προδιαγραφές, λέμε ψέματα. Διότι στην Ευρώπη θα έχουμε τον ανταγωνισμό των αμερικανικών γεωργικών προϊόντων και θα είναι πολύ σκληρός. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι γεωργοί μα. Και το λένε αυτό οι μελέτε ότι οι μικρές γεωργικέ εκμεταλλεύσεις θα είναι χαμένοι. Πρέπει να μπει στην έκθεση. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι λιγάκι αφελή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία. Οπότε έχει λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καλό θα ήταν εμείς με την γνωμοδότησή μας να επισημάνουμε τα, προβλήματα, γιατί μετά μπορεί να είναι α, κατόπιν εορτής. Ο κύριος Μπράμεν. Ο κύριος Μπράνεν. Um, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να ασχοληθώ με το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας. Η παράδοση στην Ένωση ήταν ότι εμείς αποφασίζουμε κατά πόσον ένα εισαγόμενο τρόφιμο στην Ένωση είναι ασφαλές ή όχι. Είναι κανόνα που περιλαμβάνεται στην νομοθεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, στις πρόσφατη, και στην πρόσφατη εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΤΑ. Στο TTIP, ε, ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει να γίνει τελείω αντίστροφα. Ο εξαγωγέα να είναι αυτός ο οποίος εξασφαλίζει ότι το εξαγόμενο προϊόν σέβεται τους κανόνες της ε, χώρα αγωγής. Ότι δηλαδή το Υπουργείο Γεωργίας τον είπα θα είναι αυτό που θα υλοποιεί την απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κλωμπημένων προϊόντων, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια άνευ προηγουμένου αλλαγή και δεν έχει εξηγηθεί από την Επιτροπή γιατί έγινε. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε ε, μια συμφωνία TTIP όπου τα παράστα της κάθε χώρας θα εισάγονται ελεύθερα σε, στην άλλη πλευρά δεν μπορεί οι ασθένειες των φυτών να περνούν χωρίς έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει προστασία και θα υποβάλουμε σχετική τροπολογία για να απαγορευτεί αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Νόιτσελ. Κύριε Νόιτσελ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στην Επιτροπή Γεωργίας. Άρα πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε και να αναφέρουμε τα βασικά προβλήματα για τη γεωργία. Είναι πρώτα απ' όλα αυτή η διαδικασία διαιτησίας. Και επίσης το ότι θα έχουμε μόνο ένα αρνητικό κατάλογο και όχι το θετικό κατάλογο του τι είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε διαφάνεια ούτε δημοκρατία επιπλέον. Έχουμε και γεωργικά θέματα. Για τα γεωργικά θέματα να αναφέρω τα εξή. που είναι όντω τα πιο σημαντικά το θέμα των ε, γεωργικών δομών που θα τροποποιηθούν στην Ένωση δηλαδή θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες όχι μικρότερες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υπάρξει συγκέντρωση διότι οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη ΣΥΠΑ θα δημιουργήσει συγκέντρωση και εδώ. Άρα δεν θα κερδίσουν οι γεωργοί, δεν θα αυξηθεί το γεωργικό εισόδημα και κάτι άλλο πρέπει να αναφέρουμε μια γεωργία που ε, έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η γεωργία. Εάν ε, χαιρόμεθα που καταργούνται τα εμπόδια για τις εξαγωγές μας, θα καταργηθούν και προς την άλλη κατεύθυνση τα εμπόδια. Θα βρούμε δηλαδή στις αγορές μας προϊόντα που δεν τα θέλουμε. Θα μειωθούν οι προδιαγραφές λοιπόν συνολικά και αυτό το βλέπω ιδιαίτερα επικριτικά. Ευχαριστώ κύριε Σαντριέ. Ευχαριστώ. Επιγραμματικά. Βλέπουμε ότι πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, αλλά τέτοια έκθεση έπρεπε να είχαμε κάνει και εμείς και όχι απλή γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τον κύριο Ποβέ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη γεωργία ως μεταβλητή προσαρμογής. Πρόκειται για κοινωνικό πρότυπο και θα επιμείνουμε σε αυτό. Επίσης, αν συναθεί συμφωνία τελικά, θα πρέπει να είναι συνολική, σφαιρική και ισορροπημένη για τη στρατηγική. Λάθος ε, ήταν να κάνουμε παραχωρήσεις ε, στα δοσμολογικά θέματα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είμαστε τόσο ε, υποχωρητικοί στα μη δασμολογικά. Επίσης, ε, ε, να προσέξουμε τα τελωνιακά ζητήματα στους πιο εκτεθειμένους τομείς, όπως είναι το βόλιο κρέας. Τα ευαίσθητα προϊόντα που αναφέρουν οι συγητές ε, θα πρέπει να ενημερωθούμε για το τι παραχωρήσεις έχουν γίνει, για τους μη δασμολογικούς φραγμούς, Πρόκειται για γενικέ συλλογικέ προτιμήσει ευρωπαϊκέ, δεν μπορούν να διακυβευτούν. Επίση, θέλουμε αμοιβαιότητα, δηλαδή ευθυγράμμιση και των Αμερικανικών κανόνων στι δικέ μα προδιαγραφέ. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να είμαστε πιο ε, σταθεροί και πιο αποφασιστικοί στι γεωγραφικέ ενδείξει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε του Αμερικανού να τι σέβονται μόνο όταν του βολεύει. Επίση, ε, ε, να αφαιρεθεί η παραπομπή στη συμφωνία συνολική, την οικονομική και συνολική συμφωνία με τον Καναδά, γιατί δεν νομίζω ότι είναι πρότυπο προς μίμηση. Ο κύριος Σμιθ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Από την πλευρά της πολιτικής μου ομάδας και ευρύτερα, το TTIP ξεκίνησε με λάθος τρόπο, διεξάγεται με λάθος τρόπο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει πολλά θέματα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι περισσότερο ήταν πολύ πιο αρνητική και όχι θετική. Σέβομαι τον εισηγητή, αλλά πολλοί αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα θέματα. Θέλω λοιπόν όμως να ρωτήσω τον εισηγητή μας ότι δεν θα ήταν καλύτερα και δεν θα είχε ευρύτερη συνένεση ως προσέγγιση στην Επιτροπή μας να εξαιρέσουμε το γεωργικό τομέα από το TTIP, αυτό θα βοηθήσει να ολοκληρωθεί σύντομα το TTIP, γιατί δεν είναι καλά επεξεργασμένο. Ακούσαμε ότι οι παραγωγοί μας ε, θα χάσουν ε, πολλά, ενώ δεν έχουμε επαρκή στοιχεία που να μας πείθουν ότι οι καταναλωτέ θα κερδίσουν και τόσο πολλά. Γιατί λοιπόν η Επιτροπή μας να μην κάνει μια έκκληση που να λέει ότι η γεωργία στην Ένωση δεν είναι έτοιμη για τέτοιου τύπου αντιμετώπιση. Δεν είμαστε κατά τη συζήτηση. Μπορεί να έχουμε αργότερα ε, συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, άρα να εξαιρεθεί η γεωργία από το TTIP. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, για την συζήτηση που έχουμε που δίνει σαφείς θέσεις. Άκουσα τον κύριο Νίκολσον να μιλά για σημαντικά πλονεκτήματα από τη συμφωνία αυτή. Εμένα με ανησυχεί η θέση. Η απειλή και μιλώ για την κτηνοτροφία ιδίως για το βόλιο ο κίνδυνος προκύπτει από το ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα ανοίξει στο βόρειο κρέας από τη ΣΥΠΑ. Η Συμφωνία Ελεύθερου Μπορείου μεταξύ Επιτροπής ε, και Καναδά χωρίς για 50.000 τόνους ε, συμπληρωματικούς βιοίου κρέατος ε, φτάνει τους 150.000 τόνους συνολικά δηλαδή που θα, θα εισβάλλουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα ετοιμάζουμε το TTIP με 400.000 τόνους κρέατος από τη ΣΥΠΑ. Αυτό θα είναι θα οδηγήσει για τη Γαλλία μόνο μείωση κατά 40% του εισοδήματο των ε, κτηνοτρόφων. Θα υπάρξει δε μία απειλή για την εξαιρετική παραγωγή της Γαλλίας που θα οδηγήσει σε πλήρη εξαφάνιση. Η συμφωνία αυτή δε στην ποιότητα του βορειού κρέατος είναι να δείξει ότι μια χώρα όπως η Γαλλία που έχει τις μισές ποικιλίε ζώων στον κόσμο από τις καλύτερες ποικιλίε να εξαφανιστεί προς όφελος των του, του Βορείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Κούσμιουκ, ευχαριστώ. Ελπίζω ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, δεν θα παραλυφθεί αυτό που έγινε στις διαπραγματεύσεις ε, στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Ο αρμόδιος επίτροπος τότε είχε πει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε το συμφέρον της Γεωργίας ε, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε από το εμπόριο. Δεν ελπίζω ότι στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις δεν θα έχουμε επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς. Επίσης, στα πλαίσια των ε, ευαίσθητων προϊόντων, θα ήθελα να αναβερθώ σε ένα πολωνικό ιδιαίτερα ευαίσθητο προϊόν. Τα πουλερικά. Είναι πολύ σημαντική η πτυνοτροφία και η παραγωγή αυτή ε, έχει τόσο διαφορετικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αδιανόητο και ανέφικτος ο ανταγωνισμός. Οπότε θα πρέπει να συνταχθεί ένας κατάλογος με, ευαίσθητο, με ευαίσθητα προϊόντα και μάλιστα να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα στη συμφωνία αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ κύριο Χάιταμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι η συμφωνία TTIP θα δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευκαιρία για να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και τις διατυπώσεις. Ε, πιστεύω επίσης ότι μπορούμε με το TTIP να θεσπίσουμε γενικώ πιο απαιτητικέ προδιαγραφές παντού. Οπότε και άλλη οικονομική παράγοντες θα έρθουν πιο κοντά στις δικές μας υψηλές προδιαγραφές. Όπως είπαν βέβαια και οι εισηγητές, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες ε, ισότιμου ανταγωνισμού παγκοσμίω. Με τις δικές μας ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ε, πολλοί γεωργοί χρειάζεται να κάνουν επενδύσεις για να συμμορφωθούν με αυτές. Για παράδειγμα, ε, μία απαγόρευση μιας ουσίας αύξησε το κόστος παραγωγής κατά 10%. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, η τιμή ε, για την παραγωγή σκόνης αυγού είναι 79% ε, χαμηλότερη από ό,τι αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Θα πρέπει λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Γεωργών με τις νέες συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη. Έχω μία ερώτηση ωστόσο. θα συνεχίσει να υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική που να είναι ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική διότι 30 έως 40% του ενωσιακού προπολογισμού πάνε στη γεωργία γιατί θέλουμε οι γεωργοί μας να επιβιώσουν και θέλουμε επίσης να έχουμε και προσιτά τρόφιμα, προσιτά σε τιμή. Εάν ολοκληρωθεί το TTIP θα επιβιώσει αυτού η κοινή γεωρική πολιτική. Προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος και μετά από 11 ε, έτη συμμετοχής ανακαλύψαμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες παραγωγής, συγγνώμη, οι μεγάλες αλυσίδες διανομής, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ωφελούνται κυρίως από τις εξελίξεις στο γεωρικό τομέα. Εάν λοιπόν κάνουμε, συνάψουμε το TTIP Ποιο θα συνεχίσει να παράγει προϊόντα. Τρίτον, οι προδιαγραφές, γενετικά τροποποιημένη, κλωνοποίηση, χλώριο. Βλέπουμε τι γίνεται. Θα διατηρήσουμε τις αναγκαίες προδιαγραφές για την υγεία και των καταναλωτών και των ζώων. Θα δώσουμε σαφείς απαντήσεις στους καταναλωτές μας πριν πούμε ναι σε μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Ντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βεβαίως είμαι υπέρ μιας συμφωνίας με τους Αμερικανούς, αλλά πρέπει να διατηρηθούν, να διατηρηθούν οι προδιαγραφές μας. Συμφωνώ με τον πρόεδρο του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, τον οποίο παραθέτω. Η Ευρώπη και οι Αμερικανοί πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να εισαγάγουν κοινέ προδιαγραφές που θα θέσουν το σωστό πλαίσιο για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτά λέει ο κύριος ε, Γκάμπριελ για να αποφύγουμε αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Κυρία Νόερ, λοιπόν, να μιλήσετε με τον πρόεδρο λοιπόν, του κόμματός σας. Μπορείτε μόνο να μου αναφέρετε μία περιοχή του κόσμου που να είναι πιο κοντά σε εμά από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν έχουν βεβαίω τι δικέ μα προδιαγραφέ, αλλά κανένα άλλο δεν τι προσεγγίζει τόσο πολύ, τόσο πολύ. Γι' αυτό είμαι υπέρ μια συμφωνία και νομίζω ότι ακριβώ για τα γαλακτοκομικά θα είχαμε πολλέ δυνατότητε ε, στην ε, Αμερική να πουλήσουμε τα προϊόντα μα. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι δασμοί πάνε έως 100%. Εάν καταργηθούν οι δασμοί θα έχουμε πολλές ευκαιρίες διάθεση των προϊόντων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ κύριο Παρτί, Καρτί, Μακάρθη. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τους εισηγητές για την γνωμοδότηση. Ελπίζω ότι θα δεχθούν κάποιες τροπολογίες μου, γιατί πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ με την άποψη που πολλοί φαίνεται ότι έχουν ότι εν τέλει όλα θα πάνε καλά και ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα προστατευτούν. Αν δείτε την συμφωνία από την αμερικανική οπτική και δείτε ποιοι πιέζουν τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση της ΕΠΑ για να εξασφαλίσουν την, οργάν, την λειτουργία του TTIP είναι διάφοροι εξαγωγή στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό που θέλουν είναι να μειωθούν τα επίπεδα Τις προστασίες όχι να αυξηθούν. Θέλουν να μπορούν να εξάγουν τα δικά τους προϊόντα στο δικό τους επίπεδο, κάτι που και όχι την εισαγωγή των ευρωπαϊκών προτύπων στην, στη ΣΥΠΑ. Οι προβλέψεις της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας δείχνουν ότι ε, θα αυξηθεί κατά 120% η εξαγωγή αμερικανικών προϊόντων στις, ε, στην Ευρώπη, ενώ 60% μόνο η εξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα θα μειωθεί η απόδοση των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Άκουσα διάφορους συναδέλφους να λένε ότι θεωρούν ότι είναι ευκαιρία για τη Γεωργία αυτή η συμφωνία. Χαίρομαι που σας αρέσει. Αλλά σε τι βασίζεται την άποψη αυτή. Πρέπει να τη βασίζετε σε στοιχεία. Όπως είπε ο κύριος Κάρθη. Είναι σαφέστατο. Έδωσε λεπτομέρειες ότι δεν είναι ευκαιρία. Οι μελέτες δείχνουν ότι θα θυγεί τρομερά ο τομέας του βοήου. Και θεωρώ ότι η γνωμοδότηση που θα βγάλει η Επιτροπή μας πρέπει να βασίζεται στην ε, άποψη των περισσότερων. Και έχοντας ακούσει τόσους συναδέλφους, είναι απόλυτα σαφές ότι η Επιτροπή μας ανησυχεί πολύ για το TTIP και τις επιπτώσεις του στη Γεωργία από ό,τι αναφέρει το σχέδιο γνωμοδότησης. Άρα, οπωσδήποτε, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ρωμαλαίοι και θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο από τη Σκωτία και εδώ το διπλανό μου συνάδελφο των Πρασίνων που είπαν ε, γιατί να μην εξαιρέσουμε τη Γεωργία. Η Γεωργία θα είναι απλώς ε, ένα διαπραγματευτικό ε, χαρτί το οποίο τελικά θα χάσει. Όσο και να πιστεύετε τον Άι Βασίλη, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κιόλας. Ευχαριστώ κύριε Σταραμπέλα. Δεν... Εγώ είμαι σοσιαλιστής πρόεδρος και δεν σας εκπλήσει το ότι έχω επιφυλάξεις για την συμφωνία αυτή, ιδίω στα γεωργικά ζητήματα. Δύο βασικά θέματα είναι τα σημαντικά. Πρώτον, να μην εναρμονίζουν οι δικοί τους κανόνες. Αυτό είναι αντιδημοκρατική διάλυση του συστήματος, το οποίο έχουμε κατηγορήσει. Επίσης, δεν πρέπει να μιλάμε για, δασμολογικές και, για δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια. Ε, συχνά βρίσκουμε ε, υβριστικούς ε, όρους για να αλλάξουμε κάτι. Θα πρέπει να είμαστε πιο περήφανοι για την ε, ποιότητα των προϊόντων μας και την επιστημιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ήδη αναφέρθηκε, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση της διαιτησίας στο σύστημα αυτό που ε, είναι μια επίσης προσπάθεια διάλυση του εφιστάμενου συστήματος. Ε, αυτό που επίσης πρέπει να ζητήσουμε είναι μια σαφής μελέτη που θα δείχνει, το είπε ο συνάδελφος από την Πολωνία, για τα πουλερικά. Σε κάθε χώρα υπάρχουν εκτεθειμένες παραγωγές. Αν οι εξαγωγές των ΙΠΑ προς την Ευρώπη αυξηθούν κατά 120% ενώ μόνο 60 οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τι ΗΠΑ θα υπάρξει κατάρρευση κάποιων κλάδων γιατί θα υπάρξει μια, ένας αθέμητος ανταγωνισμός που θα επιβαρύνει την ευρωπαϊκή γεωργία. Ε, το Farm Bill, για παράδειγμα, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ε, πολύ ρεαλιστικός νόμος. Δεν πρέπει να εκθέσουμε ακόμα περισσότερο τους γεωργούς μας σε ακόμα δυσκολότερες καταστάσεις από αυτές που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Σροπέ. Ε- Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να τα αναλύσουμε διεξοδικά πριν λάβουμε μια απόφαση που θα έχει σοβαρές συνέπειες. Μιλούμε για τους διάφορους κλάδους. Άλλοι θα βγουν κερδισμένοι και άλλοι χαμένοι. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες μεταξύ των κρατών μελών και τις διαφορές που υπάρχουν. Ακόμη και οι τιμές αγοράς διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μερικές τιμές είναι διπλάσιες για το ίδιο προϊόν από χώρα σε χώρα. Οπότε μερικοί τομείς ε, θα εποφεληθούν σε ορισμένες χώρες από τη συμφωνία, ενώ άλλοι θα καταβαραθρωθούν. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν ασφαλιστικές δικλείδες για να διαφυλάξουμε κάποιους τομείς ε, σε ορισμένα κρατημέλη και να αποφύγουμε ένα ντάμπινγκ των τιμών. Και κάποιοι τεράστιοι όμιλοι στις ΗΠΑ ίσως επηρεάσουν ε, τις ενεργειακές τιμές ή τις γεωργικές τιμές στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε τη γεωργία μας και τη γη μας και να βελτιώσουμε το TTIP, αντί να υπογράψουμε άρον-άρον μια συμφωνία και μετά να το μετανιώσουμε. Σας ευχαριστώ. Σάιελ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη και το συζητάμε και εδώ επί μακρόν. Έχω κάνει ε, πολλές τροπολογίες. Θέλω να πω κάτι το οποίο λείπει από μια έκθεση που θεωρώ ότι γενικά θετική. Θέλω κύριε Νίκολσον να μας πείτε ορισμένα πράγματα για την ε, κτηνοτροφία ε, που θεωρώ ότι μπορεί να έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις. Για κάποιους τομείς όμως ε, θεωρώ ότι δεν αναφέρονται στη συμφωνία. Δεν θα ωφεληθούν λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Από πλευράς Γεωργίας ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε πολύ πιο σκληρά. Γιατί αλλιώς δημιουργείται η εντύπωση ότι τα εγκαταλείπουμε όλα χωρίς να δώσουμε να πάρουμε ανταλλάγματα. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεισηγητές και εκτιμώ το πόσο μεστή είναι η γνωμοδότηση παρόλο που είναι πολύ σύντομη, μία μόνο σελίδα. Νομίζω ότι ε, έχουμε μεγάλες ευκαιρίες από την ε, συμφωνία αυτή έχουμε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα με το ρωσικό εμπάρκο. Γι' αυτό θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες ε, με τη συμφωνία αυτή για να διοχετεύσουμε τα προϊόντα μας σε άλλες αγορές. Δεν μπορούμε να λέμε βέβαια επίσης ότι τα αμερικανικά προϊόντα είναι κακής ποιότητας ενώ τα δικά μας μόνο είναι καλής ποιότητας. Απλώς θα πρέπει να θεσπίσουμε μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα και την προέλευση ζωικών προϊόντων ώστε να υποφεληθεί και ο καταναλωτής για να ξέρει τι αγοράζει στα σούπερ μάρκετ. Πιστεύω ότι η, έκθεση, ε, ότι η συμφωνία είναι υποφελής και, και θα πρέπει να την υπογράψουμε το συντομότερο δυνατό και θα λυτρώσει την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Νταντά, ο παρακαθήμενός σας. Ευχαριστώ. Παρακολουθώντας τη συζήτηση, διερωτώ με. Έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ή τώρα ξεκινάνε διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τους δύο συγητές που κατά τη γνώμη μου θέτουν καλά το πλαίσιο της συζήτησης. Αλλά πρέπει να πάμε και λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ διαφορετική ανακλάδο η κατάσταση. Αναφερθήκαμε στο κρέας, όπου υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Θα μπορούσαμε επίσης να αναφερθούμε και στον Ίνο, που θέλει να διευκρινιστούν προηγούμενες, προηγούμενες συμφωνίες μέσω αυτής της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, η Επιτροπή να μας παρουσιάσει τις απόψεις για τους τομείς που θεωρεί ευαίσθητους. Γιατί κάθε μέρα προστίθεται και άλλα ερωτήματα στο κατάλογο. Και μετά οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρχές δικαίου στην Ευρώπη. Άρα γιατί να πάμε προς ε, αυτές τις ε, ιδιωτικές δικαιοδοσίες. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο σε μια τέτοια σύμβαση. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2013 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και στην αρχή, σε Φεβρουαρίου είχαμε τον 8ο γύρο των διαπραγματεύσεων και παρατηρείται μια επίσπευση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, αυτή η διευκρίνηση. Ναι, ναι, γνωρίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει, αλλά ακούγοντα κάποια σχόλια έχω την εντύπωση ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει και έχει συναυθεί και συμφωνία. Οκ, okay, Καλώ. Η κυρία Ερά Γκαρσία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ του εισηγητές για το θετικό τόνο της ε, εργασίας τους θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία μας δίνει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Έχει πολύ δυναμικό για την Ευρώπη και για τα, ε, για τα μεσογειακά προϊόντα, οπροκυπευτικά, ε, ελαιόλαδο, ίνο. Πολλά θέματα είναι ακόμη ανοιχτά. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι η συμφωνία αυτή θα μειώσει τους κανόνες μας και ότι οι Αμερικανοί θα προσαρμοστούν σε εμά. Αμοιβαιότητα πρέπει να είναι η λέξη κλειδί και αυτή είναι η εντολή της Κομισιόν. Και μα επιβεβαιώνει ότι σε αυτήν βασίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξη για να προστατεύσει τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ε, ονομασίες προέλευση Είναι και αυτό σημείο κλειδί για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων και οπωσδήποτε Πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι τομεί που είναι ευαίσθητα προϊόντα. Τα αυγά, τα πουλερικά, τα βόια. Χρειάζονται συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Οπότε γι' αυτό θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες με βάση τη γραμμή που παρουσίασα. Πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε άλλες αγορές. Το εμπάργο της Ρωσίας ε, απέδειξε ότι είναι κορεσμένες οι δυνατότητες ε, διάθεση των προϊόντων μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε εξαγωγές για να δημιουργήσουμε και απασχόληση και γι' αυτό είναι αναγκαία η συμφωνία TTIP. Μαγκίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε δύο πολύ έμπειρους εισηγητές. Αν δείτε την πολύ σύντομη έτσι πρέπει να είναι γνωμοδότηση. Θα δείτε ότι πολλά από τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι καλύπτονται στην έκθεση. Δεύτερον, άκουσα με χαρά τον Άραν Σμιθ να κάνει το εξή σχόλιο. Δεν είμαστε αντίθετοι καταρχήν με το εμπόριο. Εγώ η Ιρλανδία είναι εμπορικό, εμπορική χώρα και έχει συμφέρον όχι μόνο για το ελεύθερο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Για το βόρειο Παρά τις ανησυχίες υπάρχουν δυνατότητες να εξαχθεί μεταποιημένο βόλιο κρέας στις ΗΠΑ όπου υπάρχουν περιορισμοί αυτή τη στιγμή. Κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν πάντα προβληματάκια και αλλαγές. Τώρα για τα, γαλακτο... για τα γαλακτοκομικά έχουμε συμφέροντα. 139% ε, δασμοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα γαλακτοκομικά προϊόντα στη ΣΥΠΑ. Να μπω λοιπόν στους συναδέλφους όπως τον κύριο Νταντά ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για μια σειρά θεμάτων. Ισοδυναμία προτύπων, για παράδειγμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τους διαπραγματευτές να προσέξουν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Η γνωμοδότηση αυτή, ωστόσο, κατά την άποψή μου, μα προχωρεί σε σημαντικό βαθμό για να καλύψει κάποια από τα θέματα που έχουμε. Και θέλω να σας ζητήσω να έχετε εμπιστοσύνη στους ε, έμπειρους διαπραγματευτές μας. Ευχαριστώ. Ο Φέντερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλή προσέγγιση στη συμφωνία TTIP που προσφέρει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά αυτό εξαρτάται από εμά αν έχουμε σωστές πολιτικές από την αρχή. Αν φοβηθούμε ότι θα μας ξεπεράσουν, θα το καταφέρουν τελικά, γιατί είναι καλύτεροι στον ανταγωνισμό. Αλλά με σωστές πολιτικές θα αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται και για την Ευρωπαϊκή Γεωργία από τη συμφωνία TTIP. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι προσέγγιση θα θετήσουμε προς τον ανταγωνισμό και την ε, αγορά μας. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά των προδιαγραφών ε, είναι το πιο ε, βάσιμο επιχείρημα κατά του TTIP. Ακόμη και αν έχουμε κοινή γεωρική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές. Διαφορετικά χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά, διαφορετικούς τρόπους παραγωγής κρέατος χρησιμοποιούμε και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά έχουμε εξασφαλίσει κάποιον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είμαι φιλελεύθερος, άκουσε την ε, Επίτροπο Μάλστρομ να λέει ότι στόχος της ΤΤΙΠ δεν είναι η υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό θα πρέπει να έχουμε συνεχώς κατά νου. Φυσικά θέλουμε ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή είναι η βάση για το τεράστιο δυναμικό ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κλάδου χάρη και στο TTIP. Σίγουρα το TTIP δεν θα μειώσει, δεν θα υποβαθμίσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαμε, εμπορικές συμφωνίες έχουμε με 50 χώρες του κόσμου. Κάθε φορά όταν ε, συνάπτουμε τις συμφωνίες θα πρέπει ε, να κάνουμε στο υπολογισμό των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων και να υπάρχει λογοδοσία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στη συγκεκριμένη συμφωνία, το TTIP. Γιατί μερικές φορές φαίνεται ότι βαδίζουμε σε ολιστηρό έδαφος. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα και να μεριμνήσουμε και για τους γεωργούς μας αλλά και για τους καταναλωτές μας έχοντας υπόψη ότι οι Αμερικανοί γεωργοί επιδοτούνται δαψιλώς και υποβοηθούνται με πολλούς και διάφορους τρόπους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τώρα θέμη τον ανταγωνισμό που ενδεχομένω δημιουργηθεί με τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν και μεταλλαγμένα στην γεωργική παραγωγή και ορμόνες και αντιβιωτικά και διαφορετικά αντιμετωπίζουν την παραγωγή τους. Οπότε οι διαπραγματευτές μας θα πρέπει ε, να τονίσουν και να διατρανώσουν τις δικές μας προδιαγραφές και τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέχρι στιγμής τέτοιες, ε, τέτοιοι κανόνες δεν έχουν, δεκτεί, ε, δεν έχουν γίνει δεκτοί από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε η χνηλασιμότητα των προϊόντων που εισάγουμε, ώστε να ξέρουν οι καταναλωτές μας τι αγοράζουν και τι τρώνε. Dziękuję pan Ευχαριστώ κύριος Πόλτσακ και μετά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και οι προσπάθειες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, Ακούστηκαν και πολλά αρνητικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε για τους Ευρωπαίους είναι σημαντική σύμμαχη σε θέματα γεωργίας. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ότι έχουν πρότυπα παρόμοια με τα δικά μας. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν ε, εξετάσεις στα διάφορα ζητήματα Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, έχουμε συμφωνίες που μπορούν να δεχθούν ανάλογες λύσεις με αυτές που Συζητούμε τώρα, άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με αντικειμενικό τρόπο. Όχι να αφήσουμε να μας ξεφύγει η ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν θετικές παράμετροι που πρέπει να καλύψουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κλάρκ, τον ε, Διευθυντή που είναι και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή πρώτα απ' όλα θέλει να ευχαριστήσει τους συζητητές γιατί θεωρούμε ότι είναι αντικειμενική η γνωμοδότηση και τους ευχαριστούμε για την ε, συντομία του κειμένου τους. Ένα σύντομο κείμενο είναι πολύ πιο πιθανό να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στο ψήφισμά της. Συμφωνούμε με τους συζητητές ότι θέλουμε να είναι φιλόδοξο αλλά πάνω απ' όλα ισορροπημένο το αποτέλεσμα στη γεωργία και πρέπει όλα τα θέματα, πρόσβαση στην αγορά, μη δασμολογική φραγμή, γεωγραφικές ενδείξεις, ε, υγειονομικά και φυτο όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Η Επιτροπή απόλυτα συμφωνεί με την άποψη των εισηγητών και πολλών μελών σήμερα ότι τίποτα που θα περιλαμβάνεται στο TTIP δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα θεμελιώδη θέματα ασφάλειας, προδιαγραφών. Δεν είναι δυνατόν να είναι πορεία προς έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή και θα αξιοποιήσουμε και την αρχή της πρόληψης. Όλα αυτά είναι σαφή και έχουν καταστεί σαφή σε κάθε επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν τα κράτη-μέλη θέλουν να εξετάσουν τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά θα δουν ότι πουθενά δεν τίθενται ένα αμφιβόλο οι προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια μέσω της συμφωνίας αυτής. Όλοι οι κανονισμοί, όλες μας οι προδιαγραφές διατηρούνται μέσω της ΕΤΑ και θα διατηρηθούν και μέσω του TTIP. Επίσης, ε, συμμεριζόμεθα τις απόψεις των εισηγητών για τα θέματα πρόσβασης στην αγορά, για τη γεωργία, η Ένωση έχει και επιθετικά και αμυντικά συμφέροντα. Πολλά μπορούμε να κερδίσουμε μέσω του TTIP στη Γεωργία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά μα, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα. Υπάρχουν ακόμη πολλοί φραγμοί όσον αφορά την πρόσβασή μα στον τομέα του κρέατο, των γαλακτοκομικών, αναφέρθηκαν. Στον τομέα του ελαιολάδου, στα ινικά προϊόντα και τα ενοπνευματόδη και τα όπορο, κυπευτικά ιδιαίτερα, τα μήλα, τα αχλάδια και τα εσπεριδοειδή. Άρα έχουμε πολλές δυνατότητε περαιτέρω Αλλά υπάρχουν και πολλές ευαισθησίε βεβαίως για ε, μερικούς ε, τομεί, Για παράδειγμα, βόιο και πουλερικά αναφέρθηκε επειδή έχουμε υψηλότερο κόστος παραγωγής, γιατί η ενέργεια είναι ακριβότερη, οι ζωοτροφές ή οι προδιαγραφές για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων συμβάλλουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί η πλήρης ε, φιλελευθερωποίηση δεν είναι εφικτή. Άρα συμφωνούμε με αυτή την έκκληση για προσοχή και σύνεση. Αναφερθήκατε σε μελέτες πολλοί ευρωβουλευτές που λένε ότι θα υπάρξει πολύ επιζήμη επίπτωση σε κάποιους ε, κλάδους της γεωργίας. Αυτές οι μελέτες όμως ε, θέτουν ως προϋπόθεση πλήρη δασμολογική κατάργηση. Βέβαια, αν υπάρξει πλήρη κατάργηση των, δεσμών, των δασμών, μπορεί να υπάρξουν αυτές οι επιπτώσεις. Πρέπει να βρούμε λοιπόν εναλλακτικέ ρυθμίσεις. Καταλήγοντας. Σημεριζόμεθα πλήρω την άποψη των εισηγητών και πολλών βουλευτών ότι μια προτεραιότητα στο TTIP θα πρέπει να είναι η καλύτερη προστασία και η εφαρμογή των ε, γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ε, επιτυχία της Ένωσης, ε, παράγονται από μικρούς παραγωγούς και μικρομεσές και επιτρέπουν στους παραγωγούς να επιτύχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Οπότε, σαφώς προτιθέμεθα να επιτύχουμε καλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως επιτύχαμε στη Συμφωνία με τον Καναδά. Και τέλος, Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με την έκκληση των εισηγητών ότι πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με πλήρως ε, διαφανή τρόπο και αφιερώντας τον αναγκαίο χρόνο. Θα το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και ο Επίτροπος ε, βεβαίως προβλέπουν στη συνεργασία με την Επιτροπή σας για το θέμα του TTIP στην περαιτέρω εξέταση του θέματος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση. Ήταν ε, πολύ καλή ανταλλαγή απόψε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η γνωμοδότηση είναι μονοσέλιδη, γιατί αυτό δικαιούμαστε μόνο. Αν ε, είχαμε τη δυνατότητα να συντάξουμε δύο δισέλιδη γνωμοδότηση θα το κάναμε. Αλλά αυτά είναι, αυτοί είναι οι κανόνες. Ο κύριος Γιάρ μας ρώτησε πριν από πολλή ώρα τι γίνεται με τα ευαίσθητα προϊόντα. Πίτερ, πολύ ευχαρίστως ε, να συζητήσουμε το θέμα των ευαίσθητων προϊόντων. Ξέρω τα πουλερικά, το βόιο κρέας, ε, τα κοτόπουλα, είναι ευαίσθητες παραγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευαίσθητα προϊόντα. Επίσης, εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, εναρμόνισης προς τα κάτω, αλλά μόνο προς τα πάνω. Μπορείτε να με θεωρείτε αφελή, αλλά ίσως ε, χρειάζεται τέτοια αφέλεια για να προωθήσουμε τα πράγματα και δεν νομίζω ότι τελικά ήμασταν αφέλεις. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα και να εθετήσουμε την πρόταση του κυρίου Σμιθ και απλώς να εξαιρέσουμε τη Γεωργία. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Δεν πρόκειται να εξαιρεθεί η Γεωργία, οπότε θα πρέπει να την υπερασπίσουμε και να τη διαφυλάξουμε καθαρά και εξάστερα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και γι' αυτό συζητούμε τη γνωμοδότηση αυτή. Και αυτή είναι η αφετηρία, όπως είπατε. Βρισκόμαστε στις αρχές. Έγιναν βέβαια συνειδητής από πέρυσι τον Ιούλιο, πρόπερση, αλλά μέχρι στιγμής γινόταν παρασκηνιακά οι συζητήσεις. Τώρα βγήκα στο φως. Τώρα ξεκινούν οι ουσιαστικές συζητήσεις και έχουμε πολύ μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Και φυσικά θα έχουμε διαφορές, ε, πεσογυρίσματα, σκαμπανεβάσματα. Αλλά φυσικά εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας είμαστε εδώ για να προτάξουμε τη θέση της Γεωργίας και να υπερασπίσουμε τους Γεωργούς μας. Σίγουρα δεν θα ικανοποιηθούμε σε όλα τα σημεία, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί να λέμε πόσο δύσκολα και πόσο απέσια θα είναι και να προκαταλαμβανόμαστε ενετικά πριν τις διαπραγματεύσεις ότι έτσι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Ευχαριστώ κύριο Δεκάστρο. Μα, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο και όσους ε, εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη δουλειά που προωθούμε ο Τζιμ και εγώ. Πολλά υπόθηκαν. Θέλω να υπογραμμίσω σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο το θέμα της διαφάνειας. Θεμελιώδες θέμα. Το υπογραμμίσαμε στο μικρό χώρο που είχαμε στη διάθεσή μας, διότι όπως θύμισε ο Τζιμ, αυτό ήταν το πλαίσιο που έπρεπε να καλύψουμε, μια σελίδα. Να υπενθυμίσω ακόμα και το λέω ενώπιον της Επιτροπής και του Διευθυντή Κλάρκ οι εμπορικέ συμφωνίες δεν τροποποιούν, δεν τροποποιούν έναν κανονισμό. Ό,τι ρυθμίζεται από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορμόνες, γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί, δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση με τι συμφωνίες. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί αλλιώ φαίνεται ότι μια εμπορική συμφωνία μπορεί να ανατρέψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω επίσης όλους τους συναδέλφους ε, συνολικά ότι μιλάμε για τις ΗΠΑ. Το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου περνά μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Δεν μιλάμε για μια μικρή χώρα, για προϊόντα, μόνο για τα γεωργικά και αγροτροφικά είναι 17 δις ευρώ ο τζίρος. Τα 5 δις ευρώ που εξάγει η Ευρώπη σε κρασί, 5 δις πέρυσι, γίνονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν γίνονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες είναι οι επιχειρήσεις που παράγουν κρασί, τυριά, λάδι, ζυμαρικά, προϊόντα που προέρχονται από τη δική μας παραγωγή, από την ε, ε, δική μας βιομηχανία τροφίμων ποιότητας που αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται. Τα τελευταία 10 χρόνια αυξήθηκε κατά 40% οι εξαγωγές προς τη ΣΥΠΑ. Δείτε και τα στοιχεία λοιπόν, συνάδελφοι. Οι μελέτες είναι σημαντικές, όλες οι αξιολογήσεις είναι αναγκαίες, γιατί το θέμα είναι λεπτό, αλλά ας δούμε και τα νούμερα. Τα τελευταία 10 χρόνια τι εξήγαγαν η ΕΠΑ προς την Ευρώπη και τι εισήγαγε η Ευρώπη από τη ΕΠΑ. Θα δείτε ότι υπάρχει ένας ενδιαφέρον χώρος που δεν θα άφηνα να ξεχαστεί. Βεβαίω, το είπαν πολλοί συνάδελφοι, είμαστε στην αρχή. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αν εμεί πούμε όχι στη συμφωνία, δεν θα υπάρξει συμφωνία αν στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα ψηφίσουμε λέγοντας συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Εμείς θέλαμε με την έκθεσή μας να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν, αλλά εγώ πιστεύω και κλείνω ότι μία θέση μας που θα είναι μόνο αμυντικού χαρακτήρα δεν είναι προς όφελος της γεωργίας στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε και μία επιθετική στάση, γιατί μιλούμε για τα συμφέροντα εκατομμυρίων εργαζομένων επιχειρηματιών στον τομέα της, ε, της γεωργίας και των τροφίμων στην Ευρώπη. Να δούμε λοιπόν και τα συμφέροντα που μπορεί να έχει η Ευρώπη από μια ε, σημαντική αγορά 350 εκατομμύρια κατοίκων με 1,5 φορά το ΑΕΠ ε, κατά κεφαλή που έχουμε εμείς. Μιλάμε για την κρίση του γάλακτος, συνάδελφοι. Τη δυσκολία του του 5% της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη που αυξήθηκε. Προς τα πού να κοιτάξουμε, ήμι μόνο στις χώρες που να κοιταξουμε η μη μονο στις χωρες που αγαπουν και θα πληρώσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ας δούμε λοιπόν με ταπεινοφροσύνη το ζήτημα, με προσοχή τα θέματα που είναι τα στάντα για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά ας δούμε και τις ευκαιρίες. Ας μην μείνουμε σε μια αμυντική στάση. Ευχαριστώ και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και οι τροπολογίες ε, λίγων οι ε, ε, προθεσμοί της τροπολογίας δίκη σε λίγες μέρες. Θα δούμε τις τροπολογίες που βάλετε με προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και θα συζητηθεί. Οπότε είναι σημαντικό να μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις μας στις πολιτικές ομάδες, προκειμένου να δημορφώσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο. Η Επιτροπή Βιομηχανίας θα ασχοληθεί με τις δημόσιες προμήθειες, με τις υπηρεσίες και άλλες επιτροπές με τις δικές τους αρμοδιότητες. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα θέματα πρόσβασης αγοράς και αυτό είναι δικό μας θέμα, γιατί θα καταργηθούν οι δασμοί. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αν θα διατηρηθεί κάποιο τμήμα, τι θα αλλάξει. Σημαντικό αυτό που είπαν ο ε, κύριος Νταντάν και η κυρία ε, Γκαρσία και τα φυτογεωνομικά θέματα και τα θέματα ε, ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικών αδείξεων. Φαντάζομαι οι δύο συνεισηγητές ε, κατέγραψαν ε, τις παρατηρήσεις και θα τις συμπεριλάβουν. Αλλά φυσικά περιοριζόμαστε στην έκταση της αγρομοδότησης. Ε, Μέχρι 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι έχετε δυνατότητα να υποβάλλετε τις προθεσμίες σας, τις τροπολογίες σας, συγγνώμη, παρακαλώ λάβετε υπόψη αυτή τη διορία. 27 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Κανονικά έπρεπε σε 11.30 να ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών, αλλά έχουμε ακόμη και το θέμα των κτηνιατρικών προϊόντων και των ιατρικών. Θα συνδυάσουμε τα σημεία 7 και 8. Μόνο γνωμοδότηση θα ετοιμάσουμε για το θέμα αυτό. Οπότε θα ακούσουμε κυρίως την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχουμε ακόμη 10 λεπτά και στις 12 παρατέταρτο θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Ο Διευθυντής παρακαλώ για την παρουσίαση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω αμέσως την, ε, τις διαφάνειες. Ελπίζω να τις βλέπετε στην οθόνη. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για αυτό το σημαντικό κανονισμό που θα είναι σημαντικός για τον κτηνοτροφικό τομέα άρα για τη γεωργία γενικότερα να σε εξηγήσω λοιπόν γιατί χρειάστηκε αυτή η αλλαγή. Οι κανόνες για την κτηνοτροφία είναι διαφορετικοί. Ανάλογα με το ποιο τομέα προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ανήγγειλε την πρόταση η διαδικασία ήταν περίπλοκη και εντατική. Η έκθεσή μας ε, ολοκληρώθηκε από μια εξωτερική εταιρεία το 2009. Είχαμε τη διαβούλευση με το κοινό το 2010. Συναντηθήκαμε μια σειρά από εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες. Είχαμε την ε, μελέτη αντικτύπου και η γνώμη η γνώμη μας ολοκληρώθηκε το 2011 και η Κομισιόν αποφάσισε επί του κειμένου αυτού το Σεπτέμβριο του 2014. Ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτόνομος κανονισμός, δεν συνοδεύεται από άλλους κανονισμούς. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή. Όλοι οι κανόνες υπογραμμίζω που έχουν να κάνουν με την κτηνιατρική περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοθέτημα. Δεν ίσχυε προηγουμένων και φυσικά θα υπάρξουν μια σειρά από εφαρμοστικές και κατοξιοδότηση πράξεις που θα έρθουν μετά. Ποια είναι τα προβλήματα δεν υπάρχουν επαρκή εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα στην Ένωση. Και υπάρχουν και προβλήματα αντιμικροβιακής αντίστασης. Αντίσταση δηλαδή στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Έχουμε επίσης ε, συγκεκριμένα τον ορισμό ποια είναι τα κύρια και ποια τα δευτερεύοντα είδη ζώων. Τα κύρια είδη ποια είναι. Είναι τα βοηδή, τα πρόβατα, τα εγωειδή, τα πουλερικά, οι σκύλοι και οι γάτες. Και τα άλλα είναι ελάσσονα. στόχο του νομοθετήματο είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των ε, κτηνιατρικών φαρμάκων για μια σειρά από είδη, σε μια σειρά από αγορές. Να μειωθεί η γραφειοκρατία, να ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Πιο πολύ σημαντικό αυτό, να ε, εισέλθουν στην αγορά περισσότερα και καλύτερα φάρμακα. και να αντιμετωπιστούν και κίνδυνοι για δημόσια υγεία όπως η αντίσταση στα αντιμικροβιακά. Ποιο είναι ο πρώτο στόχο, Αύξηση τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή συγγνώμη, θέλουμε να αυξηθούν τα κίνητρα για τον κλάδο να αναπτύξει προϊόντα ιδιαίτερα για τα ελάσσονα είδη και θέλουμε επίσης ε, να υπάρχει μία διαδικασία για ε, αδειοδότηση σε όλη την Ένωση. Και στόχος μας είναι να έχουμε τον κανόνα 10, 14 και 18 χρόνια για την αρχική έγκριση για τα κύρια είδη τα δευτερεύοντα είδη και τις μέλισσες. Αντίστοιχα, 10 για τα κύρια, 14 για τα δευτερεύοντα και 18 για τις μέλισσες. Και το θέμα της διαθεσιμότητας θα βασίσουμε την προσέγγισή μας στο να έχει σαφές πεδίο εφαρμογής το νομοθέτημα αυτό καθορίζουμε τις ε, καινοτόμες θεραπείες, ε, νέες μεθόδους, για παράδειγμα μέσω βλαστοκυτάρων και θεραπείων που βασίζονται στο αίμα. Προτείνουμε νέους κανόνες εδώ και νέους ορισμούς. Και πώς επίσης θα γίνονται οι κλινικές δοκιμές, ε, θέματα πρόβα στην αγορά και περιορισμού πρόβα στην αγορά και θέλουμε επίσης βάσει δεδομένων να είναι διαθέσιμες ε, παντού στην Ευρώπη. Και επίσης για το θέμα της γραφειοκρατίας. Υπολογίσαμε το κόστος του διοικητικού άχθους είναι περίπου 13% του, του τελικού του συνολικού κύκλου εργασιών πολύ ψηλό σε σχέση με άλλους τομείς. Όλη αυτή η διαδικασία αδειοδότησης, σήμανσης, φάρμακοεπαγρύπνησης, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Θέλουμε λοιπόν να απλουστεύσουμε τη διαδικασία. Για παράδειγμα η άδεια να είναι απεριορίστου διαρκείας, να απλοποιήσουμε τους κανόνες για τη σήμανση, την επίβλεψη, την ε, παρατήρηση των παρενεργειών. Θέλουμε επίσης να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, πολύ σημαντικό ιδίως για τις μικρότερες αγορές. Κανόνες για την επιγραμμική πώληση, η ισχύ των ε, συνταγών σε όλες τις χώρες της Ένωσης, αυτό είναι στόχος για τα φάρμακα για ανθρώπους, θέλουμε να γίνει και για τα κτηνιατρικά φάρμακα και επίσης να υπάρχουν και εθνικά συστήματα για την ε, αντίσταση στα αντιμικροβιακά. Πολύ βασικό θέμα, μια σειρά από μέτρα. Βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούνται περιορισμένα ε, τα αντιβιωτικά και ορισμένα κρίσιμα αντιβιωτικά να είναι μόνο για ανθρώπια χρήση και θα πρέπει να μην δίδεται έγκριση εάν κάποια ουσία θα μπορούσε να παίξει αρνητικό ρόλο. Ένα άλλο θέμα είναι πώς θα τροποποιείται η νομοθεσία. Θέλουμε όλοι οι κανόνες για τα κτηνιατρικά φάρμακα να είναι σε ένα νομοθέτημα για να υπάρχει ευκολότερη χρήση. Οπότε... Κάνουμε ε, μεταφορά διατάξεων άλλο κανονισμό και το δεύτερο σκέλος αφορά την λισαβονοποίηση του κανονισμού, την προσαρμογή του κανονισμού δηλαδή στην συνθήκη της Λισαβόνας. και στην ε, παρούσα δομή των κανονισμών έχουμε τον τίτλο 3 που πέρασε στον νέο κανονισμό και εκεί έχουμε πολλές διατάξεις που αφορούν τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και βλέπετε κάποια παραδείγματα διαβάζοντας προσεκτικά την πρόταση. Οι συνέπειες αφορούν την προσαρμογή του κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και μάλιστα σεβαστήκαμε γι' αυτό την ομολογία και προτείνουμε και τους κανονισμούς αλλά και κάποιες κατεξουσιοδότηση πράξεις για τις λεπτομέρειες. Κατά συνέπεια έχουμε το άρθρο 40 που αφορά την υιοθέτηση εκτελεστικών πράξεων, υπό όρους βέβαια, παρόμοιες διατάξεις χρησιμοποιήσαμε και για τον κανονισμό για την φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπους. Είχαμε αντίστοιχη διαδικασία και πέρυσι. Αυτά προσπάθησα να είμαι σύντομο. Θα επανέλθουμε στην επόμενη μας ε, παρουσίαση, στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, και μάλιστα τουλάχιστον ε, δύο φορές ακόμη γιατί η βασική συζήτηση θα γίνει τον Απρίλιο, στις 15 Απριλίου στη συνεδρίασή μας. Η σημερινή παρουσίαση έγινε για μία πρώτη εξοικείωση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γύρει προβληματισμούς, γι' αυτό και ζητήσαμε μία παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν σας ενδιαφέρει μπορούμε να σας στείλουμε και τις διαφάνειες που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχετε ένα υλικό για πιο ευρυθή μελέτη. Και το Μάρτιο, στην επόμενη μας συνεδρίαση, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με βάση τη γνωμοδότηση που θα εκπονήσουμε εμείς επί της ε, έκθεσης, της κύριης έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σήμερα δεν θα γίνει συζήτηση και ζητούμε συγγνώμη και από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τους συζητητές γιατί δεν έχουμε χρόνο για συζήτηση σήμερα. Πάντως πιστεύω ότι με την παρουσίαση απαντήθηκαν κάποιες ερωτήσεις και απορίες. Οπότε αν δεν έχετε ε, ερωτήσεις, να διακόψουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής και να περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Λυπούμε για αυτή την αλλαγή, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η παράταση της συζήτησης για το TTIP. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε λίγο και δεν προλάβαμε να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στη συζήτηση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Διακόπτουμε λοιπόν την τακτική μας συνεδρίαση και περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. is this? is Is